Okay, ladies and gentlemen, let's start. ξεκινάμε. Δεν έχει νόημα να αναμένουμε έτη περισσότερον. Σας ευχαριστώ που είσαστε παρόντες και δεν είμαι μόνος μου. Είμαστε εδώ στη δεύτερη συνεδρίαση της ημέρας. Είναι πολύ θετικό που είμαστε όλοι μαζί. <laughs> και μπορούμε να εξετάσουμε το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης Θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Λιέμα, ελπίζω σας, ε, σας ε, πρόφερα σωστά το όνομα. Είναι ο διευθυντής της ε, Μπέρεκ, που είναι ο Ευρωπαϊκός Αυτός Φορέας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και θα ήθελα να μας παρουσιάσετε την σημασία του φορέα των ρυθμιστικών, της Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνετε αποφάσεις και θα θέλαμε να ξέρουμε και κάτι για το προσωπικό σας και για τα θέματα που σας απασχολούν. Κύριε Ρέμα, σας ευχαριστώ λοιπόν που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσετε τον φορέα σας και μετά οι συνάδελφοι που παρόντες μπορούν να θέσουν ερωτήματα. And switch, I'll switch to English now, I mean, for my presentation. Θα μιλήσω αγγλικά όμως, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας τις απόψεις μου για την BEREC και την ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγομαι Άντων Ρέεμα και είμαι υποψήφιος για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στο BEREC Διευθυντή Διοίκηση στην ΠΕΡΕΚ, που είναι ο φορέα ρυθμιστικών αρχών για τι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε. Θα ξεκινήσω με μια παρουσίαση του εαυτού μου και μετά μπορείτε να θέσετε και ερωτήματα μετά. Έχω περίπου 20 χρόνια εμπειρία εργασιακή και το 1 τρίτο περίπου αυτή τη εμπειρία είναι σε άλλε χώρε και όχι τη δική μου. Και γι' αυτό ο λόγος για τον οποίο διεκδίκησα τη θέση του Διευθυντή Διοίκησης της ΜΠΕΡΕΚ ήταν πράγματι να επανέλθω κατά τα 100% σε αυτή την διεθνή αρμοδιότητα και να έχω αρμοδιότητες σε διεθνικό επίπεδο στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που καλύπτουν όλη την Ευρώπη. Έχω κάνει διοίκηση επιχειρήσεων με ένα μάστερς από ένα γνωστό Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Όπως σας είπα, έχω περίπου 20 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, περίπου 14 χρόνια ως διαχειριστής επιχειρήσεων, με ομάδες μέχρι 259 εργαζομένων και προϋπολογισμούς μέχρι 6,8 εκατομμύρια ευρώ. Είχα εμπειρία σε διάφορους τομείς εργασιακούς σε επιχειρήσεις, αλλά από το 1997 και μετά εργάζομαι ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και επίσης στην ε, βιομηχανία της, ε, των τεχνολογιών πληροφοριών. Η εμπειρία μου σε σχέση με την Μπέρεκ υπήρξε στο αξίωμα του επικεφαλής των Εθνικών Αρχών Τηλεπικοινωνιών στην ιστορία μεταξύ του 2004 και 2007. Έχω λοιπόν ποικίλε εμπειρίες, κυρίως ε, στα θέματα πωλήσεων, marketing, παροχής υπηρεσιών, που νομίζω ότι είναι σημαντικές για την BEREC, ο οποίος είναι ένας οργανισμός υποστήριξης. Το γραφείο της BEREC λοιπόν είναι ένας οργανισμός υποστήριξης και είχα την ευκαιρία να διαχειριστώ μια ομάδα η οποία υποστηρίζει τις ε, μορφές συνεργασίας για τις παγκόσμιες τηλεπικοινωνίες, ιδίως την υπηρεσία πελατών αυτού του φορέα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να έχει κανείς αυτή την εμπειρία, η οποία πιστεύω ότι είναι χρήσιμη και για την θέση του Διευθυντή Διοίκηση της ΠΕΡΕΚ. Έχω εμπειρία επίσης διαχείρισης σχεδίων σε διεθνή σχέδια με εμπλεκομένους από διάφορες χώρες και θεώρησα πάντα χρήσιμο κάθε φορά που υπάρχει ένα έργο το οποίο σχετίζεται με σχέδια να υπάρχει πάντα κάποιος με επαγγελματική εμπειρία διαχείριση σχεδίων για να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει καλά την διεξαγωγή των projects, να έχει και καλή δυνατότητα να παρέχει συμβουλές στους άλλους εμπλεκομένους. Σας είπα ποια είναι η διεθνής μου εμπειρία. Περίπου 7 χρόνια μετά και από τις σπουδές μου. 9 χρόνια συνολικά, εάν θέλετε, σε πάνω από 10 χώρες. Και το είδος, το στυλ διαχείρισής μου, πιστεύω ότι ο καλύτερος ε, διαχειριστής είναι αυτός ο οποίος μπορεί να προσαρμόζει το στυλ εργασίας του στο αντικείμενο με ένα δημοκρατικό τρόπο και με την οικοδόμηση συνένεσης, με ένα συνενετικό λοιπόν τρόπο διαχείρισης επί τη βάση των στόχων μιας επιχείρησης, επί τη βάση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται μια επιχείρηση, επί τη βάση της εμπειρίας των συναδέλφων του. και πράγματι πιστεύω ότι είναι πιο σημαντική η συνενετική διαχείριση με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας και μιας ανοιχτής κουλτούρας μέσα σε μια εταιρεία. Υπάρχουν βέβαια καταστάσεις όπου μπορεί κανείς να έχει ένα περιορισμένο προϋπολογισμό, περιορισμένο χρονικό πλαίσιο για να φέρει σε πέρα σε ένα σχέδιο, όπου δεν είναι αρκετά έμπειροι συνάδελφοι και πρέπει κανείς να έχει ένα πιο διευθυντικό στυλ. Σε πολλές περιπτώσεις προσπάθησα στην επαγγελματική μου ζωή να θέσω τα συμφέροντα του φορέα στον οποίο εργάζομαι πριν από τα δικά μου και πολλές φορές χρειάστηκα να αντιμετωπίσω στενά χρονοδιαγράμματα, κάτι το οποίο μου δίνει το κίνητρο να χρησιμοποιήσω όλες τις δυνατότητές μου και με οθεί στο μάξιμουμ της απόδοσής μου. Οι αρχές μου είναι να μεταχειρίζομαι με δίκιο τρόπο τους συναδέλφους μου, να είναι οι εκθέσεις μου βασιζόμενοι σε πραγματικά γεγονότα και να είναι οδηγοί για τη λήψη αποφάσεων, ανοιχτές επικοινωνίες και ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς στρες. Όλα αυτά λοιπόν μου δίνουν ένα λόγο να διεκδικήσω τη θέση του Διευθυντή Διοίκησης της Μπέρεκ και ως ε, διευθύνων διοίκηση στην ΠΕΡΕΚ μπορώ να φέρω την εμπειρία μου και όπως σας είπα μπορώ να δίνω κίνητρα στον εαυτό μου και να αντιμετωπίζω σφιχτά χρονοδιάγραμματα. Αυτό είναι αυτό το οποίο θέλω να κάνω για την ΠΕΡΕΚ. ως ο διοικητής της ΜΠΕΡΕΚ. Ε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε Και τώρα θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα στους αδέλφους να κάνουν ερωτήσεις, να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες. Πρώτη έχει το λόγο κύριε Τελκαστή. Ε, muchas, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για μένα είναι μια μεγάλη χαρά μια ιδιαίτερα προσωπική χαρά να συναντώ τον υποψήφιο για το Διευθυντή διοίκηση της ΜΠΕΡΕΚ. Γιατί ε, τον γνωρίζω ήδη για εννέα μήνες. Εγώ είμαι εισηγήτρια για το θέμα αυτό της ΜΠΕΡΕΚ. Ήταν δύσκολο να δημιουργηθεί η ΜΠΕΡΕΚ. Υπήρξε όλη αυτή η διαδικασία δημιουργίας και διαμόρφωσης της Μπέρεκ από την αρχική της σύλληψη μέχρι την ε, εκκίνηση αυτού του φορέα. Βέβαια υπήρξαν πολλά προβλήματα σε σχέση με το πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει αυτός ο νέος οργανισμός ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες με ένας φορέας με σημαντικές εξουσίες παρέμβασης ή ένας οργανισμός ο οποίος βασίζεται στην ήπια νομοθεσία. Δηλαδή ένας φορέας ο οποίος απλώς θα έδινε ενάσματα και θα παρακολουθούσε το έργο και της Κομισιόν και των Εθνικών Ρυθμιστών ώστε να οικοδομηθεί μια αγορά ηλεκτρών επικοινωνιών η οποία να είναι ενιαία, ανοιχτή και ανταγωνιστική γιατί αυτός είναι ο απότερος στόχος μας και τελικά γεννήθηκε η Μπέρεκ και άρχισε να μπουσουλάει κιόλα. Έχει αποφασιστεί που θα είναι η έδρα Εγώ δεν θέλω να θέσω τώρα κάποιο ερώτημα για την ΜΠΕΡΕΚ, για τις αρμοδιότητες της ΜΠΕΡΕΚ, γιατί είναι γεγονός ότι, ότι τις γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, αλλά τις γνωρίζω και εγώ πολύ καλά, διότι παρακολούθησα αυτό το θέμα. Αλλά θα έπρεπε να σας ζητήσω να πράξετε ότι είναι απαραίτητο για να γίνει η Μπέρεκ ο φορέας αυτός ο οποίος θα πρέπει να υπάρχει για μια ανταγωνιστική αγορά στις τηλεπικοινωνίες τις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες στην Ευρώπη. Για μένα το ΙΜΠΕΡΕΚ είναι ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση με τον προηγούμενο φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών που είχε απλώς το θετικό του να υπάρχει αλλά δεν υπήρχε σαφής ορισμός του έργου της ούτε το ανθρώπινο και τεχνικό υλικό. Επομένως η Μπερκ είναι ένα πολύ μεγάλο θετικό βήμα και οι αρμοδιότητες της ε, Μπέρεκ που έχουν καθοριστεί στο ρυθμιστικό τομέα της δίνουν την δυνατότητα να επηρεάσει την Κομισιόν και να της παρέχει τη δυνατότητα να επηρεάζει επίσης και τους εθνικούς ρυθμιστές. Οι εθνικοί ρυθμιστές, αυτός είναι ο απότερος στόχος, ενωμένοι σε ένα φορέα υπερεθνικού χαρακτήρα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κοιτάξουν πιο μακριά από τις εθνικές τους αγορές, από τις στενές εθνικές τους προοπτικές και να δράσουν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που έχουν ως Συμβούλιο Συμβουλευτικό και ως φορέας ο οποίος μπορεί να γνωμοδοτεί ανάλογα με τα διάφορα θέματα του επιζητούν να μπορέσουν να δράσουν μέσα σε αυτό το υπερεθνικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού πλαίσιου σε ένα τομέα ο οποίο είναι καθοριστικό για το μέλλον τη οικονομία, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και των κοινωνιών μα, και ο οποίο, πριν από ένα χρόνο όταν γεννήθηκε αυτός ο φορέας το Μπέρεκ μέσα στα πλαίσια του πακέτου των τηλεπικοινωνιών είχε να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση οικονομική όπως και όλοι μας και λόγω αυτής της οικονομικής κρίσης είναι ακόμα πιο αποφασιστικός ο ρόλος αυτού του οργανισμού γιατί ή θα προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της ψηφιακής κοινωνίας ή όλα θα χάσουν πάρα πολύ ορμή και ταχύτητα. Υπάρχουν πολλές περιοχές του κόσμου οι οποίες τώρα διεκδικούν την ηγεσία της ψηφιακής κοινωνίας είναι σαν ένα τρένο υψηλής ταχύτητος το οποίο δεν έχει κανένα σταθμό, δεν σταματάει πουθενά. Ή είναι κανείς μέσα στην ατμομηχανή αυτού του τρένου ή μένει στις ράγες του τρένου και το βλέπει να φεύγει. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι μαζί με το μηχανοδηγό. Και από την άποψη αυτή η Μπέρεκα έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Συγχαρητήρια λοιπόν, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα έχετε να αντιμετωπίσετε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο ένα έργο πρώτης τάξεως που βρίσκεται στο ύψιστο σημείο των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο να προωθηθεί η ψηφιακή ατζέντα σαν μία από τις 7 συμβολικές και εμβληματικές δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το έτος 2020 και Προφανώς εξαρτάται από σας να προωθήσετε την ΠΕΡΕΚ προς την κατεύθυνση αυτή. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία, σας εμψυχώνει η Επιτροπή μας. Εμείς θέλουμε πάντα να έχουμε συμμάχους για να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν και καλή τύχη. Ευχαριστώ κυρία Τράουτμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας άκουσα και θα σας περάσω και τις καλύτερες ευχές μου γιατί είστε ο πρώτος ε, διοικητικός υπεύθυνο ενός οργάνου το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό στην Επιτροπή μας. Με την συνάδελφο ε, Πινεύδε Καστίγιο έχετε δύο από τους τρεις σωματοφύλακες του πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες. Ο τρίτος είναι ο Μάλκομ και θα θέλαμε όλοι να δώσουμε εγγυήσει για τη λειτουργία αυτής της νέας υπηρεσίας, να της δώσουμε εγγυήσει και σχετικά με τις αρμοδιότητές της, την ανεξαρτησία της, τα νομικά της μέσα, την τοποθέτησή της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την δυνατότητα που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραμείνει, να εμπλέκεται με την υπόθεση αυτή. Είδαμε πάρα πολύ καλά πόσο η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν χρήσιμη απέναντι στους ρυθμιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι θα θέλαμε να συνεχίσουν να ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση κάποιων στρατηγικών τομέων. Το εκφράσαμε αυτό στα πλαίσια της Επιτροπής Ήτρε για την Ενέργεια, στα πλαίσια της δημιουργίας της Υπηρεσίας Ενέργειας, Ήμασταν πιο φιλόδοξοι από το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα των αποστολών που θα αναλάβει, αλλά δεν τελείωσε η διαδικασία και θα έχουμε την δυνατότητα να εκτιμήσουμε και να διατυπώσουμε νέες προτάσεις αν θεωρήσουμε ότι δεν έχουμε την δυνατότητα να επιβάλλουμε κάποια απόφαση. Για μας λοιπόν, το Μπερέκ είναι ένα μέσο το οποίο θα πρέπει να δημιουργήσει μια κάποια νομολογία στο επίπεδο της ρύθμισης του τομέα μας στην Ευρώπη, να προσδώσει εμπιστοσύνη στον τομέα αυτό σε μια κομβική στιγμή, τη στιγμή που περιμένουμε από τις επιχειρήσεις να επενδύσουν και σε επίπεδο υποδομών, αλλά και σε επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης και νέων υπηρεσιών έχετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξετε γιατί αυτό αφορά και τις ισορροπίες ανάμεσα στις χώρες μας. Έχουμε δει ότι στις διάφορες χώρες μας έχουμε ε, αποκλίνουσες απόξεις σχετικά με τις ρυθμιστικές αρχές. Το ότι θα μπορέσουμε να ομαδοποιήσουμε τις αρμοδιότητες αυτές, να τις κάνουμε να λειτουργήσουν αλληλέγγυα, να δημιουργήσουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αυτό σημαίνει ότι το ΜΠΕΡΕΚ θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και να δημιουργηθεί αυτό που είπα και πριν, μια ευρωπαϊκή νομολογία από την οποία περιμένουμε να λειτουργήσει ως είδος κινήτρου, να προσδώσει νομική ασφάλεια στις επιχειρήσεις και να επιτρέψει επίσης να ρυθμίσουμε όσο μπορούμε κάποιες συγκρούσεις με προληπτικό τρόπο και όχι πάντα σε δικαστικό επίπεδο. Αυτά σας ευχόμεθα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή η ρυθμιστική αυτή αρχή να μην έχει λόγο ύπαρξης ή τουλάχιστον όχι όπως σήμερα. Τη θελήσαμε αξιόπιστη, τη θελήσαμε ευέλικτη, εκφράζοντας τα πλαίσια αυτού του πακέτου ένα πλαίσιο αναφοράς για τον ρυθμιστή που επιτρέπει να υπάρξει σύγκληση στην συνολική αντίληψη ευθύνης αλλά και συνολική ε, ε, θα έλεγα αντίληψη πρακτικής γιατί το να είναι κανείς ρυθμιστής ε, σημαίνει ότι λειτουργεί μέσα στα πλαίσια μιας κάποιας πρακτικής. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είχαμε ήδη τη δυνατότητα να συγχαρούμε τον νέο πρόεδρο και τα μέλη. Εργαστήκαμε στενά με πολλές ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές και ωφεληθήκαμε από την συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια των εργασιών τους για τις αναθεωρήσεις των τηλεπικοινωνιών, των οδηγιών γύρω από τις τηλεπικοινωνίες. Το να αναθεωρήσει κανείς ένα τόσο σημαντικό πακέτο, ενώ έχουμε την ψηφιακή στρατηγική μπροστά μας για το 2020, σημαίνει ότι μια οδηγία ή ένα αριθμιστικό πακέτο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και να θα έλεγα γίνει αντικείμενο επεξεργασίας μαζί με αυτούς που θα το χρησιμοποιήσουν παραμένουν σε αυτή τη φάση κάποιες θα έλεγα αμφιβολίες. Παρ' όλα αυτά η διοικητική δουλειά, τα θεμέλια θα έλεγα, του Μπερέκ, εσείς θα τα αναλάβετε. Εσείς και όλοι οι συνεργάτες σας και πρέπει να γνωρίζετε ότι είμαστε πολλοί σε αυτό το κοινοβούλιο που ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Μπερέκ στα πλαίσια μια συγκυρία η οποία μερικές φορές αποκτά εκρηκτικές θα έλεγα διαστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Οπότε θα ήθελα να ξαναδώσω την ευκαιρία στον κύριο Ρήμα να μας ε, να δευτερολογήσει αν θέλει. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. περίμενα ερωτήσεις βέβαια, αλλά με βάση τις ευχές που άκουσα και την δύσκολη εντολή που έχω εγώ και η Μπέρεκ από τις ε, διακεκριμένες κυρίες εδώ πέρα. Εγώ προσωπικά θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανταποκριθώ στις ε, προσδοκίες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών οργάντων ως ε, Διοικητικός Διευθυντής, ως επικεφαλής της ομάδας μου για να ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε με ολόκληρη την ομάδα της Μάλιστα, ευχαριστώ. Ε, ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε ε, ποιες είναι οι επόμενες ε, εξελίξεις. Και με το προσωπικό, με τις... Ε, με την αποστολή σας. Εγώ δεν τα ξέρω τόσο καλά σου συνάδελφοι εδώ που είναι ειδικοί. As, mentioned, Ως υποψήφιος έχω κάνει κάποιες συζητήσεις για τους διορισμούς. Τα επόμενα βήματα είναι προσλήψεις για να αρχίσει να λειτουργεί το γραφείο και να στηθεί το γραφείο από πλευρά υποδομών, ε, βασικές ε, πολιτικές εργασίας. Έχουμε κάτι διαγωνισμό. Έχουμε δύο θέσεις ε, προκηρύξει, σημαντικές. Έχουν ξεκινήσει οι διαγωνισμοί. αναμένουμε την αξιολόγηση των αιτήσεων. Ίσως να, αυτό να γίνει το Σεπτέμβριο, βεβαίως λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Μετά έχουμε προετοιμάσει τις προκηρύξεις για α, παραπάνω θέσεις. Σε γενικέ γραμμέ, υποθέτω, α, πώς να σου το πω, στείνουμε το γραφείο στη Ρήγα τις τελευταίους μήνες του έτους και πρώτα απ' όλα ξεκινήσουμε με το διοικητικό προσωπικό αλλά μετά και τους ειδικού μάλλον στο τέλος του έτους ή αρχή του επόμενου έτους και το γραφείο θα ξεκινήσει κάποια στιγμή στην αρχή του επόμενου έτους γιατί η προθεσμία είναι τέλος Μαΐου 2011 όταν το νέο ρυθμιστικό πακέτο θα πρέπει να έχει ε, εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή αυτό για τον Μπέρεξ σημαίνει πως θα είμαστε λίγο πολύ έτοιμοι. Αυτό δεν σημαίνει πως σκοπεύουμε να προσλάβουμε όλη την ομάδα αμέσω και να περιμένουμε μετά πότε θα έρθει η δουλειά. Η δική μου η θέση είναι, και αυτό είναι και το σχέδιο, να γίνουν ε, σταδιακά τα πράγματα όσον αφορά τις ε, προσλήψεις. Και μετά να αναπτυχθεί η ομάδα όταν θα αποκτήσουμε και περισσότερο όγκο δουλειάς οι αρμοδιότητες και το στήσιμο του Μπέρεκ απαιτούν κάποια ισορροπία μεταξύ του κεντρικού γραφείου και των εμπειρογνωμόνων που θα δουλεύουν εκεί και των ειδικών που θα δουλεύουν στις εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές. Έχουμε προγραμματίσει αποσπάσεις ειδικών από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, αλλά το πού ακριβώς θα βρεθεί η ισορροπία που θα χωρίσουμε ακριβώς τη δουλειά που γίνεται. Ε, τι θα γίνει με τους αποσπασμένους ειδικού. Ε, οι λεπτομέρειες αυτές θα πρέπει ακόμα να οριστούν βεβαίως ε, και αυτό ε, θα προκύψει κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών γιατί βεβαίως και πάλι δεν μπορούμε να ε, Έχουμε πολλούς ειδικού χωρίς αυτοί οι άνθρωποι να έχουν άμεση καθημερινή ε, εμπειρία με ανάλυση της αγοράς, ε, ανάλυση ανταγωνιστικότητας ε, των αγορών ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών. Πρέπει λοιπόν να τα εξορροπήσουμε αυτά λίγο την εμπειρογνωμοσύνη εντός του γραφείου μας και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Αλλά όταν έλεγα πως το γραφείο του Μπέρεκ είναι διοικητική στήριξη για όλες τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και για το Συμβούλιο Ρυθμιστικών Αρχών. Ο στόχος της Μπέρεκ και του γραφείου αυτού θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα αποτελεσματική λειτουργία για όλους, ε, όλες τις ρυθμιστικές αρχές. γιατί θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ διοικητική δουλειά στο back office που λέμε για να μπορέσουν αυτοί οι εμπειρογνώμονες πραγματικά να κάνουν ουσιαστική δουλειά και να δώσουν ε, το μέγιστο από τη δική τους πλευρά. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κάποιος άλλος να πει τίποτα ερωτήσεις. Εάν όχι... Τότε μπορούμε να τελειώσουμε με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ τον κύριο Ρέμα. Είμαι σίγουρος πως ε, τα επόμενα χρόνια θα συναντηθούμε ούτως ή άλλως άμεσα. Εύχομαι καλή επιτυχία. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε και ήσασταν στη διάθεσή μα. Ζητώ συγγνώμη για το ότι δεν ήταν περισσότεροι συνάδελφοι εδώ πέρα σήμερα. Κρίμα. Δυστυχώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ε, είχαμε ατυχία. Εν πάση περιπτώσει σας γνωρίσαμε. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό ταξίδι. Also in die, also ich war grundsätzlich in Deutschland tätig, aber dann habe ich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 Meine Damen und Κυρίες, αγαπητοί συνάδελφοι, άλλαξαν πάλι τα θέματα στην ημερήσια διάταξη γιατί ο Ισπανός ε, Υφυπουργός ε, μας είπε ότι δεν μπορεί να έρθει γρήγορα, τελικά θα έρθει γιατί στη Γαλλία υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα. Δεν ξέρω, κυρία Τράουτμαν κάτι πρέπει να κάνει εκεί πέρα. Χαμός γίνεται με την κίνηση στη Γαλλία. Λοιπόν, το αναφέρω το επόμενο σημείο. Παρουσίαση τη μελέτη ενεργειακή αγορά ε, στον τομέα του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού, τρέχουσα κατάσταση και υλοποίηση. ορίζω τον Αντων Ρένμαλ και τον Ματίας Ατμαν. Ich, I don't know, ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen äh, startet oder wie. Ποιος θα ξεκινήσει, τι έχετε συμφωνήσει. Εγώ θα ξεκινήσω, λέει ο κύριος Άλτμαν. Σας παρακαλώ λοιπόν να μας παρουσιάσετε την μελέτη. Τώρα φοβάμαι βεβαίω ότι δεν τη διάβασαν όλοι οι συνάδελφοι, γι' αυτό σας καλέσαμε να μας τα ξαναπείτε. Παρακαλώ. Η μελέτη αυτή έχει ζητηθεί από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ήτρε το Δεκέμβριο του προηγούμενου χρόνου. Φτάσαμε μέχρι το Μάη για να κλείσουμε αυτή τη μελέτη. Και έχουμε φτάσει στην τελική μορφή λοιπόν της έκθεσης αυτής. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν, ήταν τριπλός. Καταρχήν το άνοιγμα και η συμπλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας να δούμε ποια είναι η κατάσταση του, της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού στην Ευρώπη. Δεύτερον, μια ατομιακή επισκόπηση της εφαρμογής και της μεταγραφής του δεύτερου ενεργειακού πακέτου, συζήτηση του τρίτου ενεργειακού πακέτου που πέρασε πέρσι. Το τελευταίο βήμα είναι που από στρατηγική έποψη είναι το πιο σημαντικό, είναι να αξιολογήσουμε τον δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας με τις ενδεχόμενες λακκούβες του και να προτείνουμε κινήσεις για το μέλλον. Θα σας δώσω λοιπόν μια σύντομη παρουσίαση της κατάστασης των ενεργειακών αγορών, μιλάω δηλαδή για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, και μετά θα δώσω στο συνάδελφό μου τον Άντων Ρέινχολμ για να σας δώσει περισσότερα στοιχεία για την ανάλυση των άλλων δύο πτυχών οι αγορές αυτές... Αγγλικά θα μιλήσουμε. Οι, αγγλικές, οι αγορές αυτές έχουν δύο βασικές πτυχές. Η μία είναι η φιλελευθερωποίηση και η άλλη είναι η ολοκλήρωση των αγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τη φιλελευθερωποίηση, η συγκέντρωση οικονομικών παικτών στην αγορά είναι ένας πρώτος δείκτης του τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι για την χονδρική αγορά ηλεκτρισμού. Όλες οι εθνικές αγορές στην Ευρώπη είναι σε μέτριο ή σε υψηλό βαθμό συγκεντρωμένες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε επιτύχει ορισμένα πράγματα, αλλά η εικόνα ακόμα δεν μπορεί να θεωρείται ικανοποιητική για μια απόλυτα φιλελευθερωποιημένη αγορά. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ κόκκινο ακόμα λίγο κίτρινο, λέει ο μιλητής, αλλά δεν υπάρχει στο χάρτη. Και κάποιο πράσινο, λέει πάλι ο μιλητής, που δεν υπάρχει, το οποίο δείχνει μια ιδιαίτερα υπερσυγκεντρωμένη αγορά. Αν δούμε ένα άλλο δείκτη, το πόσοι καταναλωτές αλλάζουν παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, Αυτό δείχνει όλους τους πελάτες, είτε είναι βιομηχανικοί πελάτες, είτε είναι νοικοκυριά. Και εδώ αναφέρεται το ποσοστό συνολικής ισχύω που αλλάζει πάροχο. Βλέπετε ότι και για, δεν έχουμε πληροφορίες βέβαια για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε ότι για μερικούς από αυτούς τους φορείς έχετε μηδενικό ποσοστό αλλαγής. Είναι μικρότερες χώρες και έχετε άλλες χώρες όπου το ποσοστό αλλαγής παρόχου είναι από 2 μέχρι 10, 12, ακόμα και 14 το χρόνο. Δεν είναι υψηλό ποσοστό παρόλα αυτά. Θα πρέπει να θυμόσαστε ότι αυτό αφορά τη συνολική ισχύ, τη συνολική αξία του ηλεκτρισμού, επομένως ο αριθμός των πελατών που αλλάζει είναι πολύ μικρός. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί βέβαια τώρα που είμαστε στο 2010, αλλά όχι σημαντικά η γενική εντύπωση που παίρνει κανείς από τις αγορές είναι ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό αυτό και ότι αυξάνει και η φιλελευθερωποίηση. Αν δούμε τώρα την ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έπρεπε η ολοκλήρωση να οδηγήσει σε μια ομογενοποίηση των τιμών ηλεκτρισμού σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που βλέπουμε όμως αν συγκρίνουμε πέντε σημαντικές αγορές ηλεκτρισμού είναι ότι οι τιμές δεν είναι ακόμα ενιαίες μέσα στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο μπορούμε <clears throat> να ε, διαπιστώσουμε είναι ότι οι συσχετισμοί μεταξύ των τιμών αυξάνει. Επομένως υπάρχει μεγαλύτερη κατά αυτή την έννοια σύνδεση. Αν δούμε πάλι τους δείκτες για την αγορά φυσικού αερίου, βλέπουμε ότι η συγκέντρωση στις ε, αγορές φυσικού αερίου, που είναι λιανικές αγορές για τον τελικό καταναλωτή, είναι πολύ ψηλές σε πολλές χώρες και για κάποιες χώρες μονάχα είναι μέτρια η συγκέντρωση. Αν δούμε τώρα το ποσοστό αλλαγής παρόχου για το φυσικό αέριο, και εκεί πάλι δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, αλλά στην αγορά φυσικού αερίου η φιλελευθερωπής ξεκίνησε πολύ αργότερα από ό,τι για τον ηλεκτρισμό αλλά έχει συντελεστεί με μεγαλύτερη ταχύτητα. Οπότε βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο περίπου όπως για τον ηλεκτρισμό. Και στην περίπτωση αυτή είναι <clears throat> σωστό το ότι για το φυσικό αέριο τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο 2008 και έκτοτε έχει επιταχυνθεί κάπως αυτή η διαδικασία. Τώρα, ποιες είναι οι διαφορέ μεταξύ φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Αυτό συνδέεται με την ολοκλήρωση των αγορών στην Ευρώπη. Το φυσικό αέριο εισάγεται εν γέννη το μεγαλύτερο μέρος του από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε εδώ πέρα τις εισαγωγές από την Ρωσία, τη Βόρεια Αφρική και ο τρίτος σημαντικός χώρος παραγωγής είναι βέβαια η Βόρεια Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες <clears throat> χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροφοδοτούνται από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό. Κάθε χώρα φυσικά έχει εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής. Ενώ α, βλέπουμε άρα πως η ολοκλήρωση στο επίπεδο της μεταφοράς είναι πολύ πιο προχωρημένη λόγω ακριβώ διαφοράς μεταξύ φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Από την άλλη, αυτό οδηγεί στο ότι οι χοντρικές τιμές του φυσικού αερίου είναι πολύ ε, πιο ενιαίε σε ολόκληρη την Ευρώπη από ό,τι στον ηλεκτρισμό. Και φαίνεται αυτό εδώ πέρα. Αν δείτε τη μπλε στήλη, που είναι η τιμή χοντρική σε όλα τα υπόλοιπα είναι φόροι, βλέπετε πως είναι πολύ πιο ενιαία σε σχέση με τον ηλεκτρισμό. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Αντών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ματίας και καλησπέρα σας και από εμένα. Θα εξετάσουμε λίγο την εφαρμογή του δεύτερου πακέτου και το μέλλον. Ποιε είναι οι προκλήσεις και οι συστάσεις που, θα κάνουμε. Δυστυχώ δεν έχω εγώ εικονίτσες όπως ο Ματίας. Έχω κάποιο κείμενο, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος ε, και θα τελειώσουμε στην ώρα μας. Ε, το πρώτο πράγμα προφανώς εξετάζουμε όταν εξετάζουμε την εφαρμογή του δεύτερου πακέτου είναι οι διαδικασίες ε, επί και την ένεργη, τα της ε, ενέργειας και της υποδομή στο 2009. Έχουμε πρόσβαση δηλαδή σε διασυνοριακή υποδομή, έλλειψη πληροφορίες, διαδικασίες για παράπονα καταναλωτών και ρυθμισμένες τιμές τελικού καταναλωτή. Αυτό και από τα 25 κράτη-μέλη υπάρχει ένας πίνακας που υπάρχει σελίδα 55 σχετικά. Άρα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός χωρών ε, που παραβίασαν τους κανόνες και ε, όπου δεν υπάρχουν παραβιάσεις οφείλεται στο ότι π.χ. στη Μάλτα δεν υπάρχει δίκτυο αερίου. Αλλιώς όλοι κάτι έχουν κάνει. Και τέλος έχουμε την ε, έλλειψη συστήματος ε, ποινών και φτάνουμε άρα στι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης και εδώ πέρα βλέπουμε πως οι συνήθεις εξουσίες είναι η διαφάνεια, ο ανταγωνισμός και βεβαίως η προστασία του καταναλωτή. Ο ανταγωνισμός βεβαίως είναι από κοινού με τις αρχές ανταγωνισμού, αλλά διαφέρουν σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη εξουσίες. Κάποιες εθνιστικές αρχές είναι πολύ πιο ανεξάρτητες και ισχυρές από άλλες το αναφέρουμε, θα το αντιμετωπίσουμε στο τρίτο πακέτο. Το τρίτο θέμα που εξετάζουμε είναι ο ρόλος των ε, περιφερειακών ε, πρωτοβουλειών αερίου και ηλεκτρισμού. Είναι 7 τον αριθμό, στον ηλεκτρισμό, δυστυχώς δεν έχω χάρτη και 3 στον τομέα του αερίου, οπότε διαφέρουν οι αριθμοί και αλληλεπικαλύπτονται π.χ. η Γαλλία και η Γερμανία είναι μέλη τεσσάρων διαφορετικών περιφερειακών πρωτοβουλειών οι οποίες είναι τελείως εθελοντικές και είχαμε αρκετά αποτελέσματα αλλά όπως σας είπα είναι κάτι το εθελοντικό και υπάρχει κάποια κριτική ε, βεβαίως ε, θα εξελιχθούν ακόμα είναι νέες πρωτοβουλίες ειδικά το τρίτο πακέτο θα δώσει περισσότερη ορμή αλλά η κριτική μεγαλύτερη είναι πως ε, είναι περιφερειακές ε, και ο διαχωρισμός είναι περιφερειακός και όχι λειτουργικός. Βλέπουμε πως κάποιες χώρες είναι πιο οργανωμένες στο να μοιράζονται την ε, δυνατότητα του δικτύου, οπότε θα μπορούσαν να κάνουν έναν διαφορετικό διαχωρισμό. Και το άλλο ερώτημα είναι πώς εμπλέκονται εθνικές ρυθμιστικές αρχές γιατί υπάρχει πιθανότητα κάποιες ρυθμιστικές αρχές να έχουν ελάχιστες εξουσίες το σύνολο των ε, περιφερειακών πρωτοβουλειών θα είναι ε, ο ελάχιστος ε, κοινό παρονομαστής. Γιατί αν δεν έχει κανείς αρμοδιότητες, λίγα πράγματα μπορεί να κάνει στο πλαίσιο της περιφερειακής πρωτοβουλίας και μετά έχουμε το θέμα της καθοδήγησης η καθοδήγηση δίνεται και από πάνω και πόσο, η καθοδήγηση δίνεται από κάτω προς τα πάνω. Οπότε υπάρχει μια ενδιαφέρουσα έκθεση για το τι πρέπει να, να γίνει με τις περιφερειακές πρωτοβουλίες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κομμάτι στην έκθεσή μας. Μετά περνάμε στην εφαρμογή του δεύτερου πακέτου αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το καινούριο για όσους παρακολουθούν τις αγορές της ενέργειας, πως τα μεγάλα προβλήματα αφορούν ε, τις ε, επενδύσεις και τις ενεργειακές αγορές ε, και τον προγραμματισμό. Είναι πρώτα απ' όλα η αδειοδότηση που είναι πολύ αυστηρές οι διαδικασίες. Έχουμε αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου που μπορεί να φτάσει μέχρι 7 χρόνια για τον ηλεκτρισμό. Επίσης μιλάμε για τις χρεώσεις ε, και το τι απόδοση μπορεί να έχει μία επένδυση και την ε, σταθερότητα σε βάθος 5 ή 10 ετών γιατί υπάρχουν άρα έτσι αβεβαιότητες στις επενδυτικές αποφάσεις και βεβαίως το ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται ε, επενδύσεις ε, καθώς γίνονται κάπου επενδύσεις και κάποιος άλλος κάπου αλλού εκμεταλλεύεται τα ωφέλη αυτή της επένδυσης που δεν έχει πληρώσει. Αυτά είναι στοιχεία που επηρεάζουν τις επενδύσεις. Όσον αφορά την ιδιοκτησία των συστημάτων μετάδοσης ε, και διανομής, βλέπουμε πως στον ηλεκτρισμό εξακολουθεί να υπάρχει δημόσια ιδιοκτησία από τα 26 κράτη-μέλη 18 είναι στα χέρια του δημοσίου τομέα, λιγότερο αυτό στο φυσικό αέριο, 9 από τα 24. Οπότε έχει τη μειοψηφία ο δημόσιος τομέας. Επίσης μπορεί να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας, να γύρω στο 13% όσον αφορά τον ηλεκτρισμό, αλλά μετά πάλι το πρόβλημα είναι πως οι μελέτες, ε, παρά το ότι δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς, δεν μας λένε μεμονωμένα αποτελέσματα για κάποιον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς. Οπότε δεν ξέρουμε ποιος είναι πιο αποτελεσματικός από άλλον. Όσον αφορά τη διανομή, 80% των Ευρωπαίων είναι στο καθεστώς ε, της ε, νομικής αποδέσμευσης ε, των διαχειριστών συστημάτων μετάδοσης, όπως απαιτεί νομοσία, αλλά υπάρχει και έλλειψη γνώσης, ο κόσμος δεν ξέρει πώς θα πρέπει να υπάρχει νομική αποσύνδεση του διαχειριστή του συστήματος και να είναι διακριτός και όσοι εργάζονται εκεί δεν θεωρούν πως ο διαχειριστή του συστήματος είναι αμερόληπτος. τα τεχνικές προδιαγραφές και εναρμόνιση, μας ζητήθηκε να το εξετάσουμε και αυτό και από αυτή την άποψη οι τεχνικές προδιαγραφές της ΟΚΤΕ είναι ήδη από το 2002 και δεν φαίνεται αυτό να περιορίζει την ολοκλήρωση της αγοράς στην Ευρώπη. Βεβαίως για την αιωλική η διαφορετική κωδική του δικτύου ε, μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα, αλλά οι ειδικοί λένε πως αυτό μπορεί να ξεπεραστεί. Όσον αφορά το φυσικό αέριο υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση Διευκόλυνσης Ανταλλαγής Ενέργειας, η ΕΑΣΕΕ, και ήδη από το 2002 εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση για τη ροή αερίου και υπάρχει και ένα έργο της Κομισιόν για την εναρμόνιση της ποιότητας του αερίου και υπάρχει και το site της GTE όπου φαίνονται τα διαφορά σημεία του δικτύου αερίου στην ε, Ευρώπη. Στη σελίδα 17 της έκθεσης μπορεί να βρει κανείς τον εξής πίνακα. Βλέπει κάποια από τα βασικά θέματα σχετικά με την ολοκλήρωση της αγοράς και πόσο έχει προχωρήσει κανείς στις κοινέ οργανώσεις των αγορών. Βλέπει τις διακανονισμένες τιμές, τη συγκέντρωση, για την οποία μίλησε ήδη ο Ματίας, και την λεγόμενη αποσύζευξη. Η αποδέσμευση, εν πάση περιπτώσει, είναι αυθαίρετο το ότι βάζει κανείς σε πράσινο, σε κίνητρο και σε κόκκινο. Και μπορεί κανείς όμως να διαπιστώσει ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έχουν διανύσει περισσότερη απόσταση από αυτές που έχουν μείνει πίσω. Οι μισοί τουλάχιστον Ευρωπαίοι καταναλωτές ζουν κάτω από τιμές οι οποίες έχουν περάσει από τη διαδικασία του ε, προκαθορισμού, του διακανονισμού και αυτό επηρεάζει φυσικά και τις φορολογικές πολιτικές και επηρεάζονται και οι επιδοτήσεις τιμών όπου αυτές υπάρχουν. Λοιπόν νομίζω ότι βλέπετε μία άποψη της κατάστασης. Υπάρχουν και κάποια κενά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τα δεδομένα για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως να έχει περισσότερα στοιχεία θα ήταν ίσως ιδιαίτερο κομψό για ένα οικονομολόγο να πει κανείς ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κατάλογο δικτών για το ποιος είναι πιο προχωρημένος και ποιος λιγότερο. Παρ' όλα αυτά αυτό απαιτεί περισσότερη έρευνα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει και να κάνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Σχετικά με το ποιος καθυστερεί και ποιος έχει προχωρήσει. Περνάμε τώρα στις πολιτικές του λεγόμενου τρίτου πακέτου. Έχουμε το ITO και ISO και τα διάφορα πρότυπα unbundling, αποδέσμευσης. Αυτό που βλέπουμε από τους εμπλεκομένους είναι ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ολοκλήρωσης της αγοράς μεταφοράς, δημιουργίας μεγαλύτερων μονάδων. Βλέπουμε ότι ήδη στη Γερμανία κάποιες μικρές εταιρείες έχουν πολιθεί, το ίδιο γίνεται και στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν αυτό θα οδηγήσει συστηματικά σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις με ισχυρότερη οικονομική βάση, ισχυρότεροι παίκτες δηλαδή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Υπάρχει ο κίνδυνος κάποια τμήματα αυτών των προσπαθειών στην ουσία να καλυφθούν κάτω από το άλοθη του διανομέα έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες του τρίτου πακέτου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το unbundling θέτει το ερώτημα το πόσο θα ελέγξουμε το σύστημα των διανομέων για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στο μέλλον. Η συνεργασία είναι βασικό τμήμα του τρίτου πακέτου, το ίδιο και ο προγραμματισμός των υποδομών. Οι ρυθμιστικές αρχές και και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να υπάρξει επίσης και η συνεργασία των TSO. Υπάρχει ήδη το ENSO E αγγλικά και ENSO G για το φυσικό αέριο. Όπως επίσης και τίθεται το θέμα της, ε, του προγράμματος ανάπτυξης, του δικτύου μάλλον προγραμμάτων ανάπτυξης για τα επόμενα 10 χρόνια. Ιδιαίτερα στον τομέα των ENSO E βλέπετε 28 δις για τα επόμενα 5 χρόνια να δοθούν σε υποδομές για την διανομή. Αυτό είναι μια τεράστια επένδυση η οποία απαιτείται όμως για να πάνε τα πράγματα καλά στο μέλλον. Το τρίτο πακέτο λοιπόν δημιουργεί υποχρεώσεις αλλά δίνει και ευκαιρίες για, την για τον σωστό προγραμματισμό. Θα συνεχίσω με τις πολιτικές του τρίτου πακέτου. Το θέμα είναι αν το πρότυπο στόχος, το μοντέλο στόχος θα είναι το πραγματικό μοντέλο της αγοράς στο μέλλον. Τώρα στο τρίτο πακέτο βλέπουμε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν προγράμματα στον ηλεκτρισμό τουλάχιστον για τη σύνδεση δικτύων και κατανομή δυνατότητας μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Και οι κωδικοί των δικτύων θα γίνουν δεσμευτικοί μέσω της επιτροπολογίας και θα καθορίσουν ακριβώς τους κανόνες λειτουργίας αυτού του ευρωπαϊκού μοντέλου στο μέλλον. Επίσης και το επίπεδο του εξειδικευμένου χαρακτήρα, το πώς λοιπόν θα μπορέσει κανείς να ξεκαθαρίσει τους κανόνες εκτός επιτροπολογίας έχει μεγάλη σημασία. Εν πάση περιπτώσει το τρίτο πακέτο παρέχει τις δυνατότητες για να το πετύχουμε αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί τη διαδικασία αυτή από κοντά. Οι δυνατότητες και οι αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών. Στο προηγούμενο πακέτο δεν είχαν ολοκληρωθεί. Τώρα όμως βλέπουμε ότι στα πλαίσια του τρίτου πακέτου οι ρυθμιστικές αρχές έχουν περισσότερες αρμοδιότητες έχουν περισσότερα εναρμονισμένα και αποτελεσματικά μέσα στη διάθεσή τους και θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με ευρωπαϊκό τρόπο. Το θέμα είναι το Acer που βασίζεται στη Λιουμπλιάνα, που έχει έδρα συγγνώμη στη Λιουμπλιάνα, θα είναι αρκετά ισχυρό για να λειτουργήσει σαν Ευρωπαίος ρυθμιστής. Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής θα πρέπει να εξετάσετε αν το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί εγκαίρως δεν το ξέρουμε αυτό, δεν υπάρχει μια κάποια σαφήνεια γύρω από αυτό. Αν και το δεύτερο πακέτο ή μάλλον μια και το δεύτερο πακέτο δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρω, ίσω να υπάρξουν καθυστερήσει και στο τρίτο πακέτο. Περίπου λοιπόν το έχουμε κάνει αλλά όχι εντελώ. Έχουμε προκλήσει όμω μπροστά μα. Η πρώτη πρόκληση αφορά την υποστήριξη στι ανανεώσιμε πηγέ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα και προγράμματα στήριξη των ανανεώσιμων πηγών. Επίσης και διαφορετικά νομικά πλαίσια. Αυτό δημιουργεί σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι η πιο ικανοποιητική και αποτελεσματική για την εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών. Εναρμόνιση, συντονισμός, νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να επανεξεταστούν. Υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει στα πλαίσια των μεικτών προγραμμάτων στήριξης των εναλλακτικών πηγών που έχουν προχωρήσει σκανδιναβικές χώρες. Η διαφάνεια στα οικονομικά προϊόντα, στα χρηματοδοτικά συγγνώμη προϊόντα. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες οι οποίες ρυθμίζουν τα χρηματοδοτικά μέσα εναντίον της, των καταχρήσεων από πλευράς της αγοράς και αφορά και τα ομόλογα και τις ρυθμιστικές αρχές το εμπόριο ενέργειας λοιπόν κατά κάποιο τρόπο ελέγχεται. Το θέμα είναι ποια μορφή θα πάρει αυτός ο έλεγχος και ποιο είναι ο ρυθμός με τον οποίο θα υπάρξουν συγκεκριμένε προτάσεις. Οι Ευρωπαϊκέ πολιτικές τώρα για την προώθηση ενεργειακών προγραμμάτων υποδομών και αυτό είναι κάτι το οποίο θέτει σε αμφισβήτηση αν θέλετε το ποιε είναι οι δυνατότητε που υπάρχουν για να πετύχουμε θα υπάρξει ένα πακέτο από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο τέλος ε, του 2010 και θα μιλήσουμε και για τα μέσα διασφάλισης ενέργειας ε, στο 2011. Ένας άλλος τομέας είναι οι ανταλλαγές ποσοτήτων ηλεκτρισμού. Αυτές οι ανταλλαγές ε, γίνονται κυρίως για τις εθνικές αγορές και δεν υπάρχει μια περιφερειακή διάσταση σαφής. Εδώ το θέμα το οποίο τίθεται είναι από μια έκθεση για τις περιφερειακές πρωτοβουλίες της Επιτροπής και ε, ζητείται να εξεταστεί η ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κοινού γραφείου κατανομής αυτών των ποσοτήτων. Η ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, πράγματι αυτό αφορά τις πιο ρευστές θα λέγαμε αγορές και ποιο είναι το μέλλον άραγε των συμβάσεων των μακροπρόθεσμων για τις αγορές φυσικού αερίου, τα σπότα αγορές στο μέλλον. Οι συστάσεις. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, εδώ και λίγες μέρες ε, υπάρχει συζήτηση, ε, υπήρχε συζήτηση για το τρίτο πακέτο πριν από την πλήρη εφαρμογή του δεύτερου πακέτου, οπότε είναι λογικό να συζητάμε τώρα το τέταρτο. Είναι Ήδη θα ξεκινήσει κανονικά η συζήτηση το 2011, αλλά υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις οι οποίες μπορεί να απαντηθούν. Οι ανανεώσιμες πηγές, σαν παράδειγμα. Ξέρουμε ότι έχουν κάποια προβλήματα για την πρόσβασή τους στο δίκτυο. Υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουμε τους διανομείς να προχωρήσουν στην αποδέσμευση έτσι ώστε να διευκολύνουμε την ένταξη και των ανανεώσιμων. Τι θα γίνει με τις αρμοδιότητες του Acer, είναι επαρκής και όπως είπαμε... Then again, one should remember that... των παραγόγων ε, χρειάζονται ένα αριθμιστικό πλαίσιο, αλλά δεν είναι σαν τις χρηματαγορές, δεν υπάρχει κανένα συστημικός κίνδυνος, οπότε είναι χρήσιμο να έχουμε μια αγορά παραγόγων ε, στην ενέργεια, οπότε μην το παρακάνουμε με τη ρύθμιση. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει νέες δυνατότητες. Το άρθρο 3.29 μιλάει για ενισχυμένη συνεργασία και μετά γίνονται λεπτομερείς συζητήσεις για την πρόταση Νότου Ευρώπη όπως και ο πρόεδρος ο κ. Μπούζεκ που έχει δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα και μιλάει για συντονισμό τύπου Σέγγεν, δηλαδή δίνει νέε δυνατότητε, στα κράτη-μέλη η συνθήκη. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό είναι οι επενδύσεις στην υποδομή. Βλέπουμε πως ο εναρμονισμός των συστημάτων στήριξης της Ευρώπης θα πρέπει να μας οδηγήσει σε πιο ε, αποτελεσματικά αποτελέσματα αν είναι να έχουμε ένα σούπερ δίκτυο. Πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα. Οπωσδήποτε ο προπολογισμό είναι περιορισμένο και τα ευρωπαϊκά δίκτυα για την ενέργεια δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Για να ε, κάνουμε δηλαδή μεγάλες υποδομές, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ίσως στο μέλλον να αλλάξουν τα πράγματα. Και έχουμε και το στόχο 2020-2020, σημαίνει πως πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και πώς σχετίζεται αυτό βεβαίως με την ανάγκη περαιτέρω επενδύσεων. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα δίκτυα, π.χ. φυσικού αερίου, εάν να μειώσουμε την κατανάλωση στην Ευρώπη. Αυτό ήταν ε, το δικό μας ε, το, το κομμάτι και βεβαίως να δεχτούμε ερωτήσεις ε, από τους βουλευτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χάρτμαν. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση. Βεβαίω, αν θέλουν οι συνάδελφοι να κάνουν ερωτήσει, μπορεί να το κάνουν. Πρώτα ο κύριο Ρούμπιχ ε, έχει ζητήσει τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε. Νομίζω πως είναι σημαντικό για όλους μας ε, να ξέρουμε ποια είναι η τελευταία κατάσταση της εφαρμογής. Είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την επικοινωνία σε αυτή την ε, κατεύθυνση. Είχαμε μία ψηφοφορία δε για τους μηχανισμούς εξορρόπησης ε, αντιστάθμιση μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και μια κοινή κανονιστική προσέγγιση σχετικά με την επιβολή των τελών μεταφοράς. Θα με ενδιαφέρε λοιπόν να μάθω πώς βλέπετε εσείς τον συμβιβασμό μεταξύ του κόστους μεταφοράς και της απώλειας που, έχω, που υπάρχουν όταν διέρχεται η ενέργεια από τα κράτη-μέλη. και αν θεωρείτε ότι μπορεί να καλυφθεί αυτό από το δίκτυο που κάνει την μεταφορά από πλευρά κόστου. Ευχαριστώ, κυρία Ριέρα Μαδουρέλ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω να συγχαρώ του ομιλητέ για την εργασία του και για την πολύ καλή παρουσίαση που μα κάνανε. Μα έχουν δώσει μια σειρά από δεδομένα και είναι πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα στοιχεία στο μελλοντικό μας έργο. Όλα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν να τα ακούσουμε. Όπως είπε τώρα και ο πρόεδρος, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μελετήσουμε σε βάθος τα στοιχεία της έκθεσής τους και να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό που έχει αυτή η έκθεση. Με την ευκαιρία της παρουσίας θα ήθελα να διατυπώσω μερικά ερωτήματα για τα οποία θέλω τη γνώμη σας. Καταρχήν, αναφέρατε εν τη ρήμη του λόγου αυτό το θέμα, αλλά Ποια είναι η απόψή σα για την αποκέντρωση τη αγορά φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η γνώμη σα. Δεύτερο ερώτημα. Θα ήθελα επίσης να ξέρω κατά πόσον έχετε αναλύσει τι διάφορες ρήτρε οι οποίες υπάρχουν στην εσωτερική αγορά, όπως παραδείγματο χάρη η ρήτρα τελικού προορισμού και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της αγοράς αυτής και πώς μπορούν να αρθούν ρήτες που εμποδίζουν την περαιτέρω φιλελευθερωπή της αγοράς όπως αυτές. Ευχαριστώ. Η κυρία Χέρτσοκ είχε να θέσει ένα ερώτημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ομιλητές για την εκθεσή του. Είναι πολύ σημαντικό εμείς να παρακολουθούμε όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και οι ανεξάρτητες δεξαμενές σκέψεις να παρακολουθούν τα τεκτενόμενα μετά από την εισαγωγή του δεύτερου πακέτου. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα το οποίο αναφέρεται περισσότερο στα δυνητικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούμε να προσποριστούμε. Γιατί το τρίτο πακέτο ενέργειας έχει διατυπωθεί όχι μόνο για να υπάρχει, αλλά για να προκύψουν πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές, για τους επενδυτές, για τον τομέα παραγωγής ενέργειας εν γέννη. Έχετε κάποια στοιχεία για τα πλεονεκτήματα αυτά. Επιτυγχάνουμε τους στόχους που είχαμε θέσει. Είναι το τρίτο πακέτο ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Θα πετύχουμε αυτά τα ωφέλη τα οποία αναφέραμε ή απλώς είναι πολύ ωραίο να έχουμε ευρωπαϊκές πολιτικές γραμμές. Ξέρω την απάντηση βέβαια, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποια είναι δική σας άποψη για το τι πρέπει να γίνει για να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ε, παραγωγούς ενέργειας, τους καταναλωτές και τους επενδυτές. Γιατί αυτά πρέπει να πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί αυτό είναι ο στόχος της νομοθεσίας και όχι απλώς να υπάρχει ένα πακέτο παραπάνω. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να θέσω ένα-δύο ερωτήματα. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Χέρτσοκ μας φέρνει ενώπιον του ερωτήματος για το πώς και πότε μπορούμε να αξιολογήσουμε την αναγκαιότητα ή όχι ενός τέταρτου πακέτου. Εσείς θέσατε στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής σας το θέμα της εφαρμογής. Μπορούμε λοιπόν να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα ή θα μπορούμε να ξέρουμε μονάχα όταν έχει γίνει η πλήρης εφαρμογή. Μπορούμε να έχουμε ήδη από τώρα μία τουλάχιστον εν μέρη αξιολόγηση και πώς θα μπορούμε να παρέμβουμε προτού ουσιαστικά περάσουμε στη διαδικασία του τέταρτου πακέτου, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο που θέλει το λόγο. Σα δίνω το λόγο λοιπόν. Έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε λοιπόν. Um, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την πρώτη ερώτηση δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά αλλά δεν γνωρίζω αυτές τις μελέτες. Μελέτες για τους διαχειριστές, ε, για την αποζημίωση διαχειριστών δικτύων ε, μεταφοράς ε, και διανομής. Δεν ξέρω αν έχει γίνει μια διεθνή συγκριτική μελέτη. Για την ερώτηση το, για το θέμα των πλεονεκτημάτων του τρίτου πακέτου, νομίζω αναφέραμε κάποιες πολιτικές και νομίζω πως κατά τη γνώμη μας ε, μπορούμε να δούμε πως οι πολιτικές ε, αποδέσμευσης ιδιοκτησίας, ε, προγραμματισμού των υποδομών και των κατευθυντήριων γραμμών δικτύου για να γίνουν πρώτα απ' όλα κορικοί και μετά δεσμευτικοί κανόνες είναι θετικά μέτρα του τρίτου πακέτου αλλά όπως είπα είναι δύσκολο να πούμε πριν ε, δούμε την εφαρμογή του πακέτου ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των πραγμάτων. Μπορούμε να το δούμε είτε θετικά είτε πιο επικριτικά, οπωσδήποτε. Και βεβαίω κάποιες στοιχές μπορούν να είναι καλύτερες, αλλά είμαι σίγουρος πως θα επηρεάσει τις τιμές, την ολοκλήρωση αγοράς, το πακέτο αυτό και τα λοιπά αλλά βεβαίως Κομισιόν πρέπει να φροντίσει την εφαρμογή του πακέτου. Στα κράτη-μέλη. Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το τέταρτο πακέτο, πρέπει να δούμε τι, τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη με το τρίτο πακέτο. Για τις ε, κεντρικές αγορές φυσικού αερίου και τις ρήτρε προορισμού που είπε η κυρία Ρέιρα Μαδουρέλ. Είναι δύσκολο αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν κάποια πλέον εκτήματα, αλλά... Αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ πως πρέπει να διατηρήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο μηχανισμό αγοράς γίνεται, αλλά αντιλαμβάνομαι πως αντιμετωπίζουμε μονοπόλια εκτός Ευρώπης και αυτό είναι ένα από τα... μία από τις προτάσεις που έχει γίνει. Αλλά αυτή η εξωτερική πολιτική ε, πτυχή είναι μία στην οποία δεν είμαι ειδικό και δεν θα μπορέσω να σας δώσω μία σαφή απάντηση. Ο Ματίας δεν ξέρω αν έχει να συμπληρώσει κάτι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λίγο να συμπληρώσω την κατάσταση με το φυσικό αέριο. Το θέμα είναι η αγοριστική ικανότητα. Αν συζεύξει κανείς την αγοριστική ευρωπαϊκή ικανότητα και τη στρέψει προς τις χώρες από τις οποίες εισάγει φυσικό αέριο, αυτό θα μπορούσε να επηράσει θετικά τις τιμές στην Ευρώπη. Και θα μπορούσε βέβαια να δείξει το δρόμο και σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Η Κίνα, σημαντικό παράδειγμα. Η Κίνα έχει μια τρομερή αγοραστική ικανότητα στην ενέργεια και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και με τη Ρωσία για να αγοράσουν φυσικό αέριο σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Και εκεί βρίσκεται το θέμα του πού θα πάει ο επόμενος αγωγός φυσικού αέριου προς Ανατολάς ή προς τη Δύση που λέγαμε. Μπορεί να δει κανείς ξεκάθαρα ότι η Κίνα λειτουργεί σαν μια ενιαία αγοραστική δύναμη και για τον άνθρακα. Και οι μεμονωμένοι χρήστες αντίθετα στην Δύση, οι χώρες μεμονωμένα αγοράζουν άνθρακα και έτσι έχουν μικρότερη αγοραστική ισχύ δύναμη. Αντίστοιχες καταστάσεις μπορεί να δημιουργηθούν και στην αγορά του φυσικού αερίου. Δεν υπονοώ εδώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεντρωτική αγοραστική μας ικανότητα εκεί όπου τίθεται γενικότερα το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προχωρήσω περισσότερο σε αυτόν τον τομέα. Απλά ήθελα να υπογραμμίσω λίγο τα θέματα αυτά. Ίσως με την αφορμή αυτή να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τις δύο άλλες εταιρείες και όργανα που έχουν πάρει μέρος στη μελέτη αυτή. Βλέπετε τα λογότυπα των εταιριών στις διαφάνειες μπροστά σας. Έχετε επίσης και τις διευθύνσεις μας, τις ηλεκτρονικές, είμαστε στη διάθεσή σας. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese... merci, λέει ο πρόεδρος, για τις παρουσιάσεις σας και τις απαντήσεις στα ερωτήματα. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι θέλουν να θέσουν ερωτήματα και δεν ήταν παρόντες σήμερα, πάντα έχουν τη δυνατότητα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να στείλουν ερωτήσεις για την ενεργειακή τροφοδότηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, επίσης και τους συναδέλφους οι οποίοι ήταν εδώ πέρα. Να σας ευχαριστήσω για τα στοιχεία που μας δώσανε. Οι υπόλοιποι ας διαβάσουν τα κείμενα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα της μερίσιας διάταξης. Θα περάσουν λίγα λεπτάκια μέχρι να έρθει ο προσκεκλημένος μας, αλλά έχουν έρθει εν πάση περιπτώσει. Σας περιμένουμε λίγο. So, meine Damen Λοιπόν, κύριε και κύριοι, συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Η Ισπανική Προεδρία επανήλθε. Αυτή τη φορά έχουμε τον Ισπανό Υφυπουργό Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας Πληροφορίας, τον κύριο Ρος Περάν. Είναι δύσκολο φαίνεται να έρθει κανείς σήμερα από την Ισπανία εδώ πέρα. Βεβαίω το πρόβλημα μάθαμε είναι στη Γαλλία και όχι στην Ισπανία. Όσον ήρθατε χαίρομαι που έχουμε και εκπροσώπους της Ισπανικής Προεδρίας εδώ, στις Βρυξέλλες και ε, έχουμε συνεργαστεί μαζί τους έξοχα τους τελευταίους μήνες και είχαμε καλά αποτελέσματα. Δώσαν αρκετά τώρα με τις εισαγωγές. Ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Πέραν, έχετε τον λόγο και αναμένουμε αυτά τα οποία θα μας πείτε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια μεγάλη τιμή για μένα το να τον οποίον σας για να παρουσιάσω τον απολογισμό του συνόλου των δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν προωθηθεί από την Ισπανική Προεδρία στον τομέα της ενέργειας έρευνας τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας των πληροφοριών. Είμαστε η πρώτη Προεδρία η οποία έχει ασκήσει το, την Προεδρία απολύτως κάτω από την αιγίδα της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι προσπάθειές μας είχαν σαν στόχο να ενισχυθούν και οι διαθεσμικές σχέσεις και να γίνει αποτελεσματική η τήρηση των συνθήκων στον τομέα αυτό. Συγχρόνως και με ίδια αμύωτη ένταση εργαστήκαμε για να βελτιώσουμε τις κατευθυντήριες πολιτικές γραμμές οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν και ιδίω σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο να θεσπίσουν τι απαραίτητε προποθέσει ώστε η Ευρώπη να προχωρήσει προ την εδραίωση με τι πρόοδου του τομεί αυτούς με έναν τρόπο ο οποίο θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Και φυσικά θα πρέπει να οικοδομήσουμε και τα απαραίτητα στοιχεία για να υπάρχει ένα βιώσιμο υπόδειγμα ευρωπαϊκή ανάπτυξη, το οποίο να είναι και ισορροπημένο και ανταγωνιστικό. Η επίτευξη αυτών των στόχων είναι πιο σημαντική από ό,τι ποτέ διότι είναι ακόμα ευάλωτη η ανάκαμψη και υπάρχουν οι κερδοσκοπικές επιθέσεις κατά της Ευρωζώνης που μας υποχρεώνουν να προχωρήσουμε σε βαθιές τομές, σε στρατηγικούς τομείς. Εάν η Ευρώπη <clears throat> θέλει να εξακολουθεί να είναι αυτό που ήταν στο παρελθόν, η Ήπειρος δηλαδή στην οποία συνδυάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το οικονο... η οικονομική και η κοινωνική πρόοδος θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που τίθενται ενώπιον της από τον 21ο αιώνα, ενισχύοντας τα ισχυρά της σημεία και καταπραίνοντας τα σημεία που είναι αδύνατα, για να μπορέσουμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό να επιτύχουμε το καλύτερο επίπεδο ευμάρειας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στο βαθμό του δυνατού σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό αρχίσαμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Τριάδος Προεδριών που σας παρουσιάσει ο κύριος Σεμπαστιάν στις αρχές του έτους αυτού με την βαθιά πεποίθηση ότι η ανα... ο ανακαθορισμός των πολιτικών κατά τομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας από τους κύριους φορείς της προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Μιλάω για ένα μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία πρόοδο που βασίζονται σε αποφάσεις οι οποίες έχουν αποφασιστεί σε τρεις τομείς για τους οποίους θα μιλήσω σήμερα το απόγευμα. Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και κοινωνία της πληροφορίας καθώς και βιομηχανία. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην αρχή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ενέργειας. Όπως ξέρετε, το σχέδιο δράσης για την ενέργεια, που θα πρέπει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, θα έπρεπε να είχε εγκριθεί κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Αυτό είχε ζητήσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2008, το είχε ζητήσει και το Κοινοβούλιο σας όλα αυτά. Λόγω καθυστερήσεων που επεσυνέβησαν στην έγκριση της νέας Κομισιόν, η έγκριση αυτή έχει μετατεθεί στις αρχές του 2011. <clears throat> Παρ' όλα αυτά, το σχέδιο αυτό θα υλοποιηθεί μέσα στα πλαίσια της τριάδος αυτών των προεδριών, δηλαδή της Ισπανικής και των δύο επερχομένων. Συζητήθηκε ήδη το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Ενέργειας του Μαρτίου για, το, για την προοπτική του 2020. Η Ισπανική Προεδρία πάντως θεωρεί ότι ήταν σημαντικό να δώσει στο τέλος του εξαμήνου τους ένα σημαντικό έγγραφο συμπερασμάτων για τα θέματα αυτά. Θα το εξηγήσω αργότερα και μετά από τις επαφές που είχαμε με την Κομισιόν αποφασίσαμε να συνδέσουμε το σχέδιο αυτοδράσης με την ανακοίνωση της Κομισιόν για την, για την στρατηγική της Ευρώπης 2020. Όπως ξέρετε η Κομισιόν παρουσίασε το Μάρτιο το εγγραφό τη για την νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση που περιλαμβάνει και στοιχεία σε σχέση με την ενέργεια μέσα στη στρατηγική μια Ευρώπη η οποία να είναι αποτελεσματική σε σχέση με την χρήση των πόρων. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα, η Κομισιόν παρουσίασε πρόσφατα το έγγραφο το οποίο είναι γνωστό ως ενδιάμεσο έγγραφο προς μια νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη 2011-2020 που έτυχε συζήτηση στο Συμβούλιο Υπουργών της 31ης Μαΐου μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και σε σχέση με το οποίο η Προεδρία έχει καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα τα οποία θα πρέπει να ανιβάσει για το σχέδιο δράσης στον τομέα της ενέργειας. Τα συμπεράσματα αυτά λοιπόν θα σημαίνουν επανεκκίνηση τις προσπάθειες για να κλείσει το πακέτο για τα ενεργειακά θέματα. Ένα βασικό στοιχείο αυτού του πλάνου θα είναι η ουσιαστική ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας. Για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε αυτή την ολοκλήρωση, η Ισπανική Προεδρία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε δύο βασικά στοιχεία. <clears throat> την αύξηση των διασυνδέσεων αφενός και την εναρμόνιση στο ρυθμιστικό τομέα. Για το πρώτο θέμα, για τις διασυνδέσεις, η Ισπανική Προεδρία έχει συμβάλει έντονα στην ανάπτυξη περαιτέρω διασυνδέσεων στο ενεργειακό τομέα. Συγκεκριμένα τόσο το άτυπο Συμβούλιο του Ιανουαρίου στη Σεβilla, όπως και η διάσκεψη υψηλού επίπεδου για τις υποδομές που έγινε στις 28 Μαΐου στη Μαδρίτη, έχουν δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών που θα επιτρέψουν να εγκριθεί το νέο αυτό εργαλείο για την ασφάλεια και τις υποδομές τον Νοέμβριο του 2010. Μεγάλη σημασία επίσης υπό την έποψη της προοπτικής μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας είναι και ο ρόλος <clears throat> που θα πρέπει μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας των ρυθμιστικών φορέων να παίξει η υπηρεσία ρυθμιστικών φορέων στο μέλλον. Ο φορέας αυτό θα εδράζεται στη Λουμπλιάνα, στη Σλοβενία και κατά τη διάρκεια τη Ισπανική Προεδρία δημιουργήθηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο των Ρυθμιστών και έχει διοριστεί ο διοικητή αυτού του φορέα. Σε ό,τι αφορά επίση την ασφάλεια εφοδιασμού, πέραν των δράσεων που συνάπτονται με την αύξηση των διασυνδέσεων στο ενεργειακό τομέα, θέλω να υπογραμμίσω δύο σημαντικά ακόμα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, την έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Ενεργείας της 12 Μαρτίου του 2010 του κανονισμού για την ανακοίνωση επενδύσεων σε σχέδια ενεργειακών υποδομών και δεύτερον τις εργασίες οι οποίες έχουν λάβει η χώρα ώστε το Συμβούλιο να μπορέσει να καταλήξει μια πολιτική συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση μαζί με το Κοινοβούλιο σας σε σχέση με τον κανονισμό της ενεργειακής ασφάλειας ό,τι αφορά την τροφοδοσία σε φυσικό αέριο. Όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσωρινή συμφωνία η οποία εκκρεμεί μέχρι την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πρέπει να το ψηφίσει για να το λάβει υπόψη το Συμβούλιο. <clears throat> Η Ισπανική Προεδρία θεωρεί ότι είναι ζωτική σημασία έναντι των πολιτών οι επιχειρήσεις και η κοινωνική κοινωνική σημασία φορεί να έχουν αυτά τα απαραίτητα νομοθετικά στοιχεία τα οποία εξασφαλίζουν και την ενεργειακή μα ασφάλεια. Επιπλέον, και μέσα στο πλαίσιο της ασφάλειας εφοδιασμού έχουμε παροτρύνει τον διάλογο με τρίτες χώρες. Με καταναλωτές, με παραγωγούς και με χώρες διαμετακόμισης της ενέργειας. Από την πτυχή αυτή προσπαθήσαμε να αποσύσουμε ενδεχόμενες κρίσεις εφοδιασμού για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο διατηρώντας με την Κομισιόν τους απαραίτητους μηχανισμούς έγκαιρης προεδοποίησης και παρακολούθησης που θα αποφύγουν την επανάληψη καταστάσεων όπως αυτές που ζήσαμε στο παρελθόν. Στην πρόσφατη δοκιμασία που έχουμε ζήσει τις τελευταίες μέρες, Ευτυχώ λειτουργήσε καλά αυτό ο μηχανισμό όπω ξέρετε. Επίση, σε σχέση με τι εξωτερικέ μα σχέσει, θέλω να τονίσω την εφαρμογή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου τη Ισπανική Προεδρία ομάδων εργασίας διατλαντικού χαρακτήρα, τη ομάδα εργασίας διατλαντικού χαρακτήρα για την ενέργεια μαζί με τι Ηνωμένε Πολιτείες. Και αυτή η ομάδα εργασία θα συνεχίσει να εργάζεται κάτω από φλαμαντική προεδρία. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κάνουμε τι απαραίτητε ενέργειες για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα τη ασφάλεια ενέργεια, τη αποδοτικότητα ενέργεια και των ανανεωσίμων ενεργειών. Η Σουηδική Προεδρία ήδη παρουσίασε το 2006 ένα σχέδιο για την ενημέρωση στους τομείς αυτούς, αλλά αυτή η πρόταση που ε, έγινε επί Σουηδικής Προεδρίας δεν έχει οδήσει ακόμα σε πρόταση από την πλευρά της Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά, η Ισπανική Προεδρία, όπως είναι λογικό, θεωρεί ότι θα πρέπει μέσα στο σχέδιο δράσης για την ενέργεια να συμπεριληφθεί και αυτή η πρόταση σαν τμήμα ενός αδιάσπαστου συνόλου η Ισπανική Προεδρία μπόρεσε να περατώσει εργασίες της Σουηδικής Προεδρίας σε ό,τι αφορά τα θέματα της, ε, της ε, αποδοτικότητας των κτίριων, ενεργειακής αποδοτικότητας και της ε, ετικέτας ενεργειακής απόδοσης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η νομοθεσία για, την ενεργή, για τις εναλλακτικές ενέργειες πριν από ένα έτος, αλλά θεωρούμε ότι είναι υψίστης σημασία η μεταγραφή της στις εθνικές νομοθεσίες και από την άποψη αυτή εργαστήκαμε για να προωθήσουμε την εφαρμογή των σχεδίων εθνικής δράσης που θα πρέπει να υποβάλλονται στην προσοχή της Κομισιόν μέχρι τις 31 Ιουνίου. Λόγω της αβεβαιότητας σε σχέση με τις πτυχές αυτής της οδηγίας, ιδίως ό,τι αφορά τις, τα θέματα συνεργασίας, θέλω να τονίσω τη σημασία του σεμιναρίου για την ε, τι ανανεώσιμε ενέργειε που είναι στην Παμπλώνα 15 και 16 Απριλίου. Ήταν ο καταλληλότερο χώρο για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να προετοιμάσουν τα αντίστοιχα του εθνικά σχέδια. Μέσω τη ε, κοινή διατύπωση μια φιλόδοξη πολιτική για τι ανανεώσιμε ενέργειε που περιλαμβάνει σαφεί στόχου και επίση αποτελέσματα στο οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Καταβάλαμε προσπάθειε στον τομέα τη ενεργειακή τεχνολογία για μια οικονομία χωρίς άνθρακα, όπως λέει και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, χωρίς την τεχνολογία οι στόχοι μας σε σχέση με την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή δεν θα είναι πραγματοποιήσιμη. Η Ισπανική Προεδρία γνωρίζει πολύ καλά αυτή τη σημαντική διάσταση για την ενεργειακή μας πολιτική, επίσης και για την πολιτική απασχόληση και βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες στον τομέα αυτό. Επί τη βάση να επενδύσουμε στο μέλλον των τεχνολογιών χαμηλής χρήση άνθρακος που ενεκρίθη από την Κομισιόν τον Οκτώβριο του 2009, η Ισπανική Προεδρία ε, κατέληξε σε μια σειρά συμπερασμάτων που μετά από την αντίστοιχη διαδικασία συζήτησης ενεκρίθησαν και από το Συμβούλιο Ενέργειας της 2 της Δευτέρας Ματίου. Τα συμπεράσματα αυτά έχουν σε στόχο να συμβάλλουν στην εκκίνηση πρωτοβουλειών σε βιομηχανικό επίπεδο που θα επιτρέψουν την περαιτέρω πρόοδο για τις πηγές καθαρής ενέργειας. Συμπληρωματικά με τα συμπεράσματα αυτά έλαβε χώρα και η διάσκεψη κορυφής του λεγόμενου SET Plan 3 και 4 Ιουνίου και μετά από την οποία ξεκίνησαν επίσημα από τους βιομηχανικούς φορείς οι τέσσερις πρώτες πρωτοβουλίες μεταξύ των επτά πρωτοβουλειών που έχουν θεσπιστεί σε βιομηχανικό επίπεδο, δηλαδή αιωλική ενέργεια, αιωλική ενέργεια, εφή δίκτυα και ε, δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακος ο Υπουργό κ. Σεμπαστιάν ε, όταν εμφανίστηκε ενώπιον σα για να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας αναφέρθηκε στα θέματα αυτά συγκεκριμένα. Στο παρελθόν η ενέργεια από ορυκτά καύσιμα ήταν αιτία πολέμων και συγκρούσεων. Γιατί ήταν πάντα κάτι που εποφθαλμιούσαν τα διάφορα κράτη για οικονομικούς λόγους και αυτό οδηγούσε σε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Είναι καιρό να ξεπεράσουμε κάτι τέτοιο με τις ανανεώσιμες ενέργειες οι οποίες είναι ανεξάντλητες και καθαρές δίνει τη δυνατότητα βιωσιμότητας και συνεργασίας και ειρήνης κάτι το οποίο εμείς ως Ευρωπαίοι δεν μπορούμε παρά να το εκμεταλλευτούμε. Αυτό είναι το πνεύμα το οποίο μας οδήγησε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Ισπανικής Προεδρίας να προωθήσουμε μεταξύ άλλων το σχέδιο για την ηλιακή ενέργεια στη Μεσόγειο ως μία από τις προτεραιότητες του εξαμήνου μας. Στις 11 και 12 Μαΐου στη Βαλένθια κάναμε μια διάσκεψη σε σχέση το σχέδιο αυτό, το Plan Solar Mediterráneo, για να αντιμετωπίσουμε μαζί με τους βιομηχανικούς φορείς και τις, τους χρηματοοικονομικούς φορείς τα σύνολα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Τα συμπεράσματα της διάσκεψης της Βαλένθια θα <clears throat> έλθουν στην επόμενη Υπουργική Διάσκεψη ε, της Ευρώπης της, ε, της Ένωσης για τη Μεσόγειο που θα γίνουν το επόμενο καλοκαίρι. Και επομένως έτσι θα προχωρήσει το σχέδιο αυτό για την ηλιακή ενέργεια στη Μεσόγειο. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο έλεγχος της ενέργειας είναι και θα είναι και στο μέλλον ένα κομβικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αλλά δεν είναι το μόνο τέτοιο στοιχείο οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας αποτελούν ένα άλλο σημαντικό φορέα ανάπτυξης και ενοτομίας και ανταγωνιστικότητος και θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε και τώρα και στο μέλλον για να μπορέσουμε να εξακολουθούμε να διεκδικούμε την οικονομική, τεχνολογική ηγεσία και την ηγεσία στον τομέα των υπηρεσιών σε παγκοσμίο επίπεδο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι έτσι και γι' αυτό το λόγο η πρώτη πρωτοβουλία της ε, Ισπανικής Προεδρίας στον τομέα αυτό ήταν η σύγκληση προς, η πρόσκληση μάλλον προς τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες ε, τηλεπικοινωνιών για να διατυπώσουν τις βασικές τους μέρημνες ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να ενισχύσει και να διευρύνει ακόμα περισσότερο τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τις υπηρεσίες στον τομέα της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών. Στις 18 Ιανουαρίου οι ευρωπαϊκοί φορείς ε, τεχνολογίες των Πληροφόρων και επικοινωνιών παρουσιάσανε στην Ισπανική Προεδρία <clears throat> τις θέσεις τους σε σχέση με μια συνολική στρατηγική. Το έγγραφο αυτό περιλάμβανε ένα σύνολο από προτάσεις τις οποίες έχει αναδιατυπώσει η Ισπανική Προεδρία προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, τα μέσα ενημέρωση για να υπάρξει και λήψη υπόψη των μέσα στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας 2010-2015. Η Ισπανία θέσπισε σαν μία από τις βασικές προτεραιότητές της το ότι η ψηφιακή ατζέντα 2010-2015 να εγκριθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου Ισπανικής Προεδρίας και γι' αυτό έχουμε κρατήσει μια στενή και μόνιμη επαφή με τους φορείς της Κομισιόν που είναι επιφορτισμένοι με την επεξεργασία της νέας αυτής στρατηγικής. Συγχρόνως έχουμε συμβάλει στην, στον καθορισμό των κυρίων οδηγών γραμμών που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ψηφιακή ατζέντα. Στις αρχές του έτους διατυπώσαμε μια ισπανική πρόοδο πρόταση μάλλον την ε, στρατηγική της Γρανάδας που είναι η θέση της Ισπανικής Προεδρίας για τα θέματα αυτά που διατυπώθηκε και προς τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του 2010. Αυτή η πρόταση ζητούσε η Ευρώπη να ενισχύσει τις προσπάθειές της και να προωθήσει περισσότερο την κοινωνία των πληροφοριών στο χρονικό διάστημα 2010-2015 θέτοντας τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές στο επίκεντρο της ψηφιακής επανάστασης. Και Τονίζοντα ότι αυτή πρέπει να είναι η ραχοκοκαλιά των προσπαθειών της Ισπανική Προεδρίας για την ισότητα και την καινοτομία. Τονίστηκε επίση η σημασία του να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στον ψηφιακό περίγυρο μέσα από την έγκριση μιας χάρτας δικαιωμάτων των καταναλωτών και χρηστών στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας. Εξάλλου, επειδή γνωρίζουμε ότι αυτές είναι οι τεχνολογίες οι οποίες είναι γεωγραφικά οικουμενικές στη φύση τους και οι οποίες θα γίνουν απόλυτα οικουμενικές σε ό,τι αφορά την κατανάλωσή τους, ήταν απαραίτητο να ενισχύσουμε και τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών. Έλαβε χώρα μια πρώτη συνάντηση τον Ιανουάριο στην Ουάσιγκτον με τους εκπροσώπους της Αμερικανικής κυβέρνησης με τους οποίους αντιλάχισαν ιδέες και σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης και μετά από τέσσερα χρόνια, χωρίς να έχει γίνει μια τέτοια εκδήλωση, υπήρξε μια άλλη σημαντική εκδήλωση που οργανώθηκε από την Ισπανική Προεδρία και ήταν η σύγκληση του 5ου Υπουργικού Φόρουμ Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής 14 και 15 ε, του Μαρτίου στην Γκράνχα κοντά στη Μαδρίτη με το σύνθημα ψηφιακό περιεχόμενο για μια ψηφιακή κοινωνία. Μέσα στο φόρμα αυτό υπήρξε ένα απολογισμό των δημοσίων πολιτικών για τι πολι... τεχνολογίε και επικοινωνία για την ψηφιακή ατζέντα με του κοινου στόχου, να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα και να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη μέσω τη συνεργασία. αλλά λαμβάνοντα πάντα υπόψη τι ιδιαιτερότητε κάθε περιοχή. Και ω εκ τούτου οι παρούσε χώρε, όπω και η Περιφερειακή Φορή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΘΕΠΑΛ που είναι η Οικονομική Επιτροπή για την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική εξάλλου υπογράψαμε μια κοινή δήλωση της Γκράνχα που περιλαμβάνει μια σειρά ιδεών και αρχών ξεκινώντας από την αναγνώριση της αξίας των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε ό,τι αφορά την, τα ευφυή συστήματα μεταφοράς ενέργειας και των ε, μεταφορών μπορούν να προωθήσουν τον κοινό αυτό στόχο. Αυτά ήταν και τα στοιχεία στη συζήτησή μας στην άτυπη συνεδρίαση που έγινε στις 17 ε, Απριλίου στη Γρανάδα. Η Ισπανική Προεδρία παρουσίασε ορισμένε πολιτικές θέσεις οι οποίες κατέληξαν στην ομόφωνη έγκριση από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της λεγόμενης δήλωση της Γρανάδα για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα. Η δήλωση αυτή περιείχε τους κύριους άξονες οι οποίοι είναι απαράγραπτοι για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πραγματική οικονομία και κοινωνία ψηφιακή που να είναι καινοτόμα και περιεκτική. Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 5 Μαΐου του 2010 το ψήφισμα, <clears throat> ένα ψήφισμα σε σχέση με μια νέα ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη 2010-2015 και το Μάιο επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη, μια ανακοίνωση όπου προέτεινε μια Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα για το 2010-2015 και αυτό ήταν ο πρώτος από τους βασικούς άξονες Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, ο οποίος υλοποιείται με αυτόν τον τρόπο, περιλαμβάνοντας ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνει νομοθετικά μέτρα και ειδικέ δράσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να εξέλθουμε από την κρίση και να προετοιμάσουμε την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επερχόμενη δεκαετία. Αυτή η ατζέντα περιλαμβάνει και την χάραξη μιας οδού για τη μεγιστοποίηση της ε, επιρροής των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, ιδίως για την διεύρυνση των δυνατοτήτων ευρυζωνικών επικοινωνιών στο ίντερνετ και με στόχο να βελτιωθεί η οικονομική δραστηριότητα και η καθημερινή ζωή και των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στον πρόλογο αυτή τη ψηφιακή ατζέντα λέγεται ότι οι δράσει αυτέ οι οποίε προτείνονται στου διάφορου τομεί οι οποίοι έχουν εντοπιστεί βασίζονται σε διαβουλεύσει με διάφορου εμπλεκόμενου και επίσης στα πλαίσια της δήλωσης της Γρανάδας και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει λοιπόν όλων αυτών των στοιχείων, το, το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 31 Μαΐου υπεστήριξε την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα και την διαβίβασε προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο έλαβε χώρα στις 17 Ιουνίου υποστηρίζοντας ένα φιλόδοξο σχέδιο με δύο βασικές πτυχές. Αφενός, δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, ιδίω των μικρών και μεσαίων, και επίσης την έγκριση συντονισμένων ε, μέτρων για τη βελτίωση των δικτύων, της ασφάλειας και της συγχωρητικότητας των δικτύων για να προωθηθεί ακόμα περισσότερο η χρήση του και η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων καταναλωτών και των χρηστών στον κυβερνόχωρο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης στην συνεδρίασή του της 17ης Ιουνίου απεφάσισε, παραθέτω, μετά από την παρουσίαση από την πλευρά της Κομισιόν της πρώτης αυτής πρωτοβουλίας ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει τη δημιουργία αυτού του φιλόδοξου προγράμματος, το οποίο θα βασίζεται σε συγκεκριμένες προτάσεις και παρακινεί και παροτρύνει όλους τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεσμευτούν να το εφαρμόσουν πλήρως και μέχρι κεραίας μεταξύ των του οποίου να περιλαμβάνεται και η δημιουργία μιας ψηφιακής οικονομίας αγοράς μέχρι το 2015, πέρα της παράθεσης. Εάν γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά, η ψηφιακή ατζέντα θα μας οδηγήσει σε μια ψηφιακή οικονομία μέσα στην οποία θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητες των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλους τους τομείς και έτσι να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε καλύτερα τις παγκόσμιες και συνολικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα προς μια οικονομία που θα είναι πιο αποτελεσματική σε ό,τι αφορά τη μικρότερη χρήση ενέργειας. Κλείνουν λοιπόν σε σχέση με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, θέλω να αναφερθώ σε άλλες τρεις τεχνικές συνεδριάσεις που έγιναν κάτω από την αιγίδα της Ισπανικής Προεδρίας. Μία για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στο ίντερνετ, όπου ενεκρίτη μια συμφωνία η οποία θέτει τις βάσεις συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτόν τον τόσο σημαντικό τομέα. Επίσης μια δεύτερη συνεδρίαση σε σχέση με την ηλεκτρονική υπογραφή που προώθησε σημαντικά τον εντοπισμό των απαραίτητων μέτρων για την προώθηση αυτής της σημαντικής πρακτικής που θα πρέπει να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις ε, αποτελεσματικότητας και μείωση κόστους και τρίτον μια ακόμα πιο σημαντική ίσως ε, συνεδρίαση για την χρήση μετρικών και τη λήψη αποφάσεων στην ε, κοινωνία των πληροφοριών με παρουσία της Διεθνούς Ένωσης Τηλεοπικοινωνιών ενεκρή τη συμφωνία της ε, Μαδρίτης που θέτει τις βάσεις για εξυγχρονισμό και παρακολούθηση των παραμέτρων και των μοντέλων για τις μετρήσεις και τους δείκτες στον δυναμικό αυτοτομέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Τόσο το μοντέλο αυτό λοιπόν το ενεργειακό όσο και η χρήση των προαναφερθέντων τεχνολογικών είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για να μπορέσουμε να προωθήσουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία του μέλλοντο. Χωρί όμω ένα ισχυρό και εύρωστο βιομηχανικό τομέα δεν θα μπορεί να υπάρξει αυτή η κοινωνία. Κυρίε και κύριοι, όπω είπε και ενώπιον τη Επιτροπή σα ο Υπουργό κ. Σεμπαστιάν, η οικονομική κρίση είχε τεράστιο αντίκτυπο στη βιομηχανική δράση όλων των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω εκ τούτου, ετέθησαν εν κινήσει σε πολλά κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρα υποστήριξη προς τον βιομηχανικό τομέα. Είναι απαραίτητο να σκεφτούμε περισσότερο σε σχέση με την καταναλωτικότητα αυτών των μέτρων και να προωθήσουμε μια συζήτηση σε σχέση με την αναγκαιότητα μιας νέας πολιτικής βιομηχανικού επίπεδου με τον ορίζοντα του 20 και του 20. Μέσα σε όλα αυτά, το Συμβούλιο της 1ης Μαρτίου, το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, ενέκρινε μια σειρά από συμπεράσματα σε σχέση με τις προτεραιότητες της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκαλών την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατυπώσει μια νέα ανακοίνωση για τη βιομηχανική πολιτική μέχρι το τέλος του 2010. Θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική θα πρέπει να σε θέση να υποστηρίξει την βιωσιμότητα και την καινοτομική δυνατότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για να μπορέσει να εξασφαλίσει και την αγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η όθηση λοιπόν προς την βιωσιμότητα και την καινοτομικότητα, όπως πρέπει να πω πέντε μήνες Υπουργό κ. Σεμπαστιάν, είχε μέσα από την αυτοκινητοβιομηχανία ένα από τους καλύτερους συμμάχους του μέσω του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για το βιομηχανικό μέλλον το οποίο θα προωθηθεί μέσα από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά πρόκειται και για το ενεργειακό μέλλον μας και το τεχνολογικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να στοιχηματίσουμε στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο σημαίνει ότι ενσωματώνουμε τις ανανεώσιμες ενέργειες στον τομέα των μεταφορών, μειώνοντας την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο. Η Ισπανική Προεδρία λοιπόν το έθεσε αυτό στα κέντρο, στο κέντρο τη ε, ατζέντα τη για να μπορέσουμε να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα συγκεκριμένα το πετρέλαιο και να μειώσουμε τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακο για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια για να βελτιστοποιήσουμε την καμπύλη ζήτηση του ηλεκτρισμού. Όλα αυτά λοιπόν θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στο να ξανατοποθετήσουμε σε ηγετική θέση την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία μετά από την οικονομική κρίση και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από πετρέλαιο και να προωθήσουμε την εξοικονόμηση και την πιο ορθολογική χρήση της ενέργειας και δίνοντας τη δυνατότητα να υπάρξει ένα ποιοτικό άλμα σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες ενέργειες υπέρ και του περιβάλλοντος. Επίσης και από τεχνολογική άποψη, επειδή το ηλεκτρικό αυτοκίνητο σημαίνει και την ε, ανάπτυξη λογισμικού και επίσης τεχνολογιών ε, συσσωρευτών και ευφυά και ξύπνια δίκτυα είναι πολύ σημαντικό και η Ισπανική Προεδρία θέλει να προωθήσει μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τα ενδεχόμενα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λεφθούν για να προωθηθεί η χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία και να προωθήσει τη μεγαλύτερη χρήση του στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό τον λόγο στο άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα του, Σαν Σεμπαστιάν τον Φεβρουάριο μιλήσαμε για το μέλλον του ηλεκτρικού αυτοκινητού στην Ευρώπη. Η εμπλουτιστική συζήτηση στην Τονόστια έδειξε ότι τα κράτη-μέλη συμμερίζονται κάθε ενδιαφέρον για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και είναι πεπισμένες για το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει το αυτοκίνητο αυτό το ηλεκτρικό για την αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης. Είναι σαφές ότι ορισμένε χώρε θέλουν μια ανοιχτή στρατηγική, μια ευρέως φάσματος τεχνολογική δυνατότητα, άλλοι όμως θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ω αποτέλεσμα αυτή τη συζήτηση, 28 Απριλίου, η Κομισιόν παρουσίασε ένα, μια ανακοίνωση σε σχέση με τα καθαρά αυτοκίνητα και την ενεργειακή τους απόδοση και επίσης 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα όπου ζητούσε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η παρουσία του ηλεκτρικού αυτοκίνητου. Τρίτον, στις 25 Μαΐου το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ενέκρινε μία σειρά συμπερασμάτων στις οποίες υπεστήριζε τη θέση της Κομισιόν σε σχέση με την εφαρμογή όλων των μέτρων υποστήριξης προς τα καθαρά αυτοκίνητα που περιλαμβανόταν στο σχέδιο δράση Ως εκ τούτου, η Ισπανική Πρόεδρια κατέβαλε πολύ μεγάλε προσπάθειε να προωθήσει μια κοινή στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ω εκ τούτου είναι σαφέ ότι χρειάζονται περαιτέρω πρόοδοι στον τομέα αυτό για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μαζί με τις κυβέρνησεις Πορτογαλίας, Γαλλίας και Γερμανίας υπεγράφει μια κοινή δήλωση για την πρόθεση του ηλεκτρικού αυτοκίνητου στην Ήπειρό μας. Εξάλλου, στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής, η Ισπανική Προεδρία είχε σαν στόχο να ενισχύσει το, την πρόθεση του λεγόμενου A Small Business Act. Και να μπορέσει λοιπόν <clears throat> αυτό το νομοθέτημα για τις μικρές επιχειρήσεις να προωθήσει την βελτιστοποίηση των κοινών πρακτικών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο ήταν αντικείμενο ενός συνεδρίου στη Μαδρίτη 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Εν ώψη της επικείμενης μεταρρύθμισης του νομοθετήματο για τι μικρέ επιχειρήσει, η Κομισιόν θέλει να το συνδέσει με τη στρατηγική του, της Ευρώπης 2020 και έχει διαπιστώσει ότι οι κατευθυντές γραμμές δράση τη θα πρέπει να κατευθυνθούν προ την κατεύθυνση τη καινοτομία τη επιχειρηματική αύξηση της εξέβρεσης χρηματοδότησης, της διεθνοποίησης και της προώθησης στην ψηφιακή ατζέντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και εξάλλου, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του εξαμήνου της Ισπανικής Προεδρίας, θέλω να υπενθυμίσω την πολιτική συμφωνία η οποία εξέβρεται σε σχέση με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, βάσει της οποίας εξασφαλίζονται εναρμονισμένες συνθήκες για την εμπορία των προϊόντων κατασκευαστικού χαρακτήρα. Και επίσης τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα, 25 Μαου σε σχέση με τη μελλοντική ε, μεταρρύθμιση του συστήματος σημάτων. Θα κλείσω κυρίες και κύριοι. Η Ευρώπη βρίσκεται στο πιο σημαντικό και υπερβατικό ίσως στοιχείο της ιστορίας της. Από τότε που ξεκίνησε σαν ένα ευρύ σχέδιο αλληλεγγύης μεταξύ χωρών με κοινέ πολιτικής. Η πιο ολέθρια κρίση στον οικονομικό τομέα των τελευταίων ετών με σημαντικέ αρνητικές συνέπειε σε παγκόσμιο επίπεδο και κερδοσκοπικέ επιθέσεις μας υποχρεώνουν να προχωρήσουμε σε βαθύε τομές οι οποίε θα ενισχύσουν και τη δυνατότητα τη Ευρώπη, και αυτό θα δοκιμάσει την ικανότητα των θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κατασκευάζουμε, να οικοδομούμε την Ευρώπη από την Ευρώπη και προ την Ευρώπη. Η Ισπανική Προεδρία εργάστηκε λοιπόν όλο αυτό το εξάμεινο αόκνος με μόνο μία ιδέα. Μόνο με περισσότερη Ευρώπη μπορούμε να έχουμε μέλλον και στον τομέα των, των τομεακών πολιτικών ο στόχος μας είναι να συνενώσουμε, να μην διχάσουμε και να συνεχίσουμε μια προσπάθεια βιώσιμη και ε, μόνιμη η οποία θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενώπιών μας, προκλήσεις για τις οποίες θα πρέπει τώρα να αναλάβει τη σκητάλη η Προεδρία και στην οποία ευχόμαστε κάθε επιτυχία για να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το σημαντικό έργο, το οποίο δεν είναι μόνο δικό μας, αλλά είναι το έργο όλων των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υφυπουργέ. Μετά τις πολύ λεπτομερείς ε, εξηγήσεις σας έχουμε τώρα δυνατότητα να θέσουμε και ερωτήσεις. Έχουμε λοιπόν Κάποιοι αδέλφους. Η κυρία Ρέιρα Μαδουρέλ θα ξεκινήσει. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να α, καλωσορίσω τον κύριο Υπουργό, τον ευχαριστούμε για την παρουσία του και θα ήθελα να τον συγχαρώ και για την εργασία την οποία έχει επιτελέσει τους τελευταίους μήνες ε, γύρω από τα θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του. Έχουν πετύχει αρκετά πράγματα σε πολλούς περίπλοκους τομείς θα έλεγα που μας ενδιαφέρουν και εμάς. Η Ισπανική Προεδρία μπόρεσε να εργαστεί με εντατικό τρόπο καταθέτοντας το πρόγραμμά της στην αρχή της Προεδρίας από τον Υπουργό Σεμπαστιάν, ένα πρόγραμμα πάρα πολύ φιλόδοξο και βλέπουμε τώρα με ικανοποίηση ότι το πρόγραμμα αυτό εν πολλής έχει ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολό του. Μας δώσατε πολύ ξεκάθαρες ε, εξηγήσεις για τις προσπάθειες που έγιναν τους τελευταίους έξι μήνες. Δεν υπάρχουν πάρα πολλέ ερωτήσει γιατί οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι ικανοποιητικέ. Θα ήθελα να κάνω εδώ τώρα μια αναφορά σε μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας. Αυτό το οποίο εσείς υπογραμμίσατε σαν βασικό στόχο στα πλαίσια των οδικών μεταφορών ήταν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που είπατε ότι ήταν μια σαφής εναλλακτική λύση. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα καθαρά αυτοκίνητα, τα οποία εξοικονομούν επίσης ενέργεια, προέβλεπε μια ολόκληρη σειρά από συγκεκριμένες δράσεις γύρω από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και εμείς υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα και εσείς αναφερθήκατε και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Υπάρχει κάτι όμως το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί. Πιστεύετε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να περιμένουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει την διατύπωση των μέτρων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα δράσης ή πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κατάλληλο πλαίσιο έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να αναπτύξουν τα εθνικά τους προγράμματα υποστήριξης στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μια δεύτερη ερώτηση γύρω από το ίδιο πάντα θέμα. Στα πλαίσια της δυνατότητας του ύπαρξης των διαφόρων εθνικών πολιτικών, ποιες είναι οι προσδοκίες οι οποίες υπάρχουν σχετικά με τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λειτουργήσει συντονιστικά. Από όλα αυτά τα μέτρα αυτό που έχει σημασία είναι να λειτουργήσει σωστά η εσωτερική αγορά. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν ποια από τα μέτρα τα οποία αναφέρατε πιστεύετε ότι είναι τέτοιου είδους τα οποία θα πρέπει να ενεργοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Πριν κλείσω όμως θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από πολλούς συναδέλφους, όχι μόνο της πολιτικής μου ομάδας, αλλά και από άλλες πολιτικές ομάδες, οι οποίοι λόγω ημέρας και ωραρίου ζητούν συγγνώμη. Και η κυρία Καστίγιο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δυστυχώς έπρεπε να αποχωρήσει. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μπαντία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κύριο Υφυπουργό που ήρθε εδώ πέρα. Ευχαριστώ την Ισπανική Προεδρία που έρχεται τόσο συχνά στην Επιτροπή μας και παρουσιάζει το πρόγραμμά της Σήμερα λοιπόν κάνουμε αυτόν τον απολογισμό. Με συγχωρείτε που έλειπα πριν, ήμουν στην Επιτροπή Απολιτισμού με την Υπουργό Παιδείας, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα από την Ισπανική Προεδρία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε. Όπως ξέρετε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ασφάλεια των προμηθειών, ενέργειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Τι άποψη έχετε, έχει γίνει κάποια πρόοδος επί ε, Ισπανικής Προεδρίας. Πώς αξιολογείται αυτό το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας. Ευχαριστώ. Κλοντ Τούρμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ήδη είπα σήμερα το πρωί στον συνάδελφό σας από την Ισπανική κυβέρνηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισπανική κυβέρνηση που σε μια τέτοια περίοδο κρίσης συνέχισε να αναλαμβάνει τις ευθύνες της γύρω από την Προεδρία. Ο κατάλογος των δραστηριοτήτων σας στον τομέα της ενέργειας και της βιομηχανίας είναι σαφώς εντυπωσιακός το ότι μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την οδηγία γύρω από την ασφάλεια και για το φυσικό αέριο νομίζω ότι οφείλεται και σε εσά. και της κυρίας Μπεατρής Συνεβάς, η οποία πραγματικά μας βοήθησε να οδηγήσουμε σε θετικά αποτελέσματα τις προσπάθειές μας. Και αυτό αναγνωρίστηκε από όλους εδώ στο Κοινοβούλιο και οι προσπάθειες σας στις ανανεώσιμες ε, πηγές και η συνάντηση στην Παμπλώνα και η συνάντηση στην Βαλένθια για τη Μεσόγειο. Εν θα μπορούσα να συνεχίσω οι προσπάθειες τις οποίες κάνετε σαν παράδειγμα για την προώθηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ε, γύρω από, τα, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δείχνει ότι έχουμε μια προεδρία που δεν έχει μόνο οράματα αλλά είναι μια προεδρία η οποία σταδιακά προσπαθεί να αντιθέσει σε λειτουργία αυτή τη στρατηγική και αυτά τα οράματα. Πέρα από αυτή την παρένθεση θα ήθελα να πω ότι είναι κρίμα που καθυστερήσατε και πρέπει να συζητήσουμε εδώ ε, με πολύ λίγο κόσμο παρόντες, αλλά οι βουλευτές οι οποίοι είναι παρόντες παρακολούθησαν προσεκτικά τις εργασίες σας και εκτιμούν την προσπάθειά σας. Η ερώτησή μου, η πρώτη μου ερώτηση, αφορά την προσπάθεια που κάνατε για τη Μεσόγειο θάλασσα. Είμαι σχετικά διστακτικός εγώ σε σχέση με αυτό που ονομάζω μεγάλες πολιτικές γιορτές της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Ας είμαστε ειλικρινεί, όσο υπάρχει το πρόβλημα ανάμεσα στο Ισραήλ και η Παλαιστίνη και δεν πρόκειται να διαλυθεί το πρόβλημα αυτό σύντομα, έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη γιορτή θα έλεγα, η οποία όμως δεν προχωράει ουσιαστικά. Το μήνυμά μου στην συνάντηση της Βαλένσια ήταν ότι μάλλον αυτό που χρειάζεται είναι να εντοπίσουμε σωστά δύο-τρεις από τις χώρες της Μεσογείου που έχουν ανανεώσιμα προγράμματα όπως η Τινησία, η Αίγυπτος, ε, το Μαρόκο το οποίο έχει την δυνατότητα να συνδέεται ήδη ηλεκτρικά με την Ισπανία και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα μέτρα διμερή έτσι ώστε να προχωρήσει το πρόγραμμα ηλιακής ενέργειας για τη Μεσόγειο. Φοβάμαι ότι αν παραμείνουμε πάντα σε επίπεδο όπως ονομάζεται μεταπολιτικής δεν θα προχωρήσουμε. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τη διασταύρωση ανάμεσα στις πολιτικές ενέργειας και τις βιομηχανικές πολιτικές. Γνωρίζω ότι στη χώρα σας έχει υπάρξει μια κάποια πολεμική που ξεκίνησε από τη μελέτη ενός κάποιου καθηγητή πανεπιστημίου στη Μαδρίτη, ο οποίος είπε ότι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας είναι κάτι που καταστρέφει θέσεις απασχόλησης στην ισπανική οικονομία. Διάβασα τη μελέτη αυτή, εξεπλάγην, δεν τη βρίσκω πάρα πολύ σοβαρή σε επίπεδο επιχειρηματολογίας και επιστημονικής επάρκειας. Εσείς που είστε υπουργός, εσείς που με άλλους στην Ισπανία συνοδεύσατε όλες αυτές τις επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών. Τι αποτελέσματα έχουν δώσει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τώρα που συζητάμε την βιομηχανική πολιτική να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η Ευρώπη να βγει από την κρίση και πώς μπορεί η Ευρώπη να επαναβιομηχανοποιηθεί και εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει μέσα από τις πράσινες τεχνολογίες. Δώστε μας λοιπόν πληροφορίες για το τι συμβαίνει στον τομέα αυτό στην Ισπανία. Κυρία Χέρτσογκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό που ήρθε εδώ. Εμένα μου άρεσε πάντα όταν συναντούσαμε τους υπουργούς στο τέλος του εξαμήνου, γιατί τότε κάνουμε απολογισμό και είναι κρίμα το ότι ασχοληθήκατε κυρίως με την οικονομική κρίση και τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών και έτσι επισκιάστηκαν τα αποτελέσματα και η πολλή δουλειά που έχετε κάνει. Οπότε είναι χρήσιμο το ότι ήρθατε σήμερα εδώ πέρα και μας υπενθυμίσατε αυτά τα πράγματα που ξέρουμε, αλλά επισκιάζονται από την κρίση. Όπως το ΙΣΕΡ, ψηφιακή ατζέντα, η διάσκεψη περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είχα έρθει και εγώ στο Σαν Σεμπαστιάν και είδα πως ε, επηρεάζονται οι ισπανικές επιχείρησεις. Ως δε ε, Ουγγαρέζα, μακάρι η Ουγγρική Προεδρία να έχει ένα τέταρτο της δικής σας δραστηριότητας. Θα είναι φοβερή επιτυχία. Τέλος μία ερώτηση έχω μόνο. Πώς βλέπετε τη βιομηχανική πολιτική, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την ψηφιακή ατζέντα να δένουν έτσι για να προωθηθεί ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εάν συνδεθούν αυτές οι πολιτικές θα έχουμε ένα αποτέλεσμα έτσι, θετικό. Ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα και είστε μαζί μας, με όσοι είμαστε εδώ, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ, Παύλο Ρουμπίχη. Και εγώ να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε χρόνο να έρθετε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί νομίζω πως η Ισπανική Προεδρία ε, έχει καταφέρει κάποια πράγματα σημαντικά για εμάς, όπως παραδείγματος χάρη υπόψη για τον Μπέρεκ και η απόφαση επιτέλους να ξεκινήσει να λειτουργεί το Μπέρεκ είναι πολύ σημαντικό για την ε, τεχνολογία αυτή της επικοινωνιών και της πληροφορικής και καλό θα είναι το Μπέρεκ να υποστηριχθεί πρώτα απ' όλα στους, ε, να υποστηριχθούν οι εθνικοί πρωταθλητές ε, και να πάνε στις υπόλοιπε 26 αγορές. Δηλαδή να, η κυρίαρχη εταιρεία στην κάθε χώρα να εμφανιστεί ως νέα εταιρεία στις υπόλοιπε 26 αγορές για να υπάρξουν έτσι και νέοι κορυφαίοι παίκτες και βεβαίως η εκπροσώπηση των καταναλωτών μας από τις εθνικές χώρες της 26. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία έτσι ώστε οι πολίτες μας και οι βιομηχανίες μας, οι υπόλοιπες 26 χώρες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες όπως γίνεται αυτό στην ε, μητρική αγορά της κάθε μίας εταιρείας. Ένα ερώτημα τώρα, το οποίο είναι σημαντικό για τους πολίτες μας στην Ευρώπη, είναι το roaming δεδομένων, η περιαγωγή δεδομένων. Έχουμε τώρα πάρα πολλά έξυπνα τηλέφωνα όπως λέγονται και ε, κατεβάζουν πάρα πολλά δεδομένα ή πολίτες ε, ε, και με ταχύτητες που είναι μέχρι 100 Mbps. Αν το μετατρέψουμε αυτό σε τιμές, έχουμε στόχο 50 λεπτά του ευρώ ανά Μbps. Αυτό σημαίνει δηλαδή 50 ευρώ το λεπτό με αυτή την ταχύτητα. Οπότε πρέπει να προειδοποιήσουμε λίγο τον κόσμο εδώ πέρα. Δεν θεωρείτε λοιπόν πως με τη νέα αυτή μορφή επικοινωνίας θα έπρεπε να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην τους γδίνουν εδώ τους καταναλωτές αλλά να υπάρχει έτσι, περισσότερη διαφάνεια για να μην έχουμε έτσι, κατάχρηση αυτής της ώρας. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Να ζητήσω λοιπόν από τον κύριο Υπουργό να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Bien, eh, muchas gracias. Mil merci, λέει ο Υπουργός. Πρώτα απ' όλα, Θέλω εκ βάθους καρδίας να ευχαριστήσω εξ ονόματος της Ισπανικής Προεδρίας, εξ ονόματος όλων μας που έχουμε εργαστεί τόσο έντονα αυτό το εξάμεινο, ώστε παρά την κρίση και παρά τις καθυστερήσεις που επεσυνέβησαν για την ενθρόνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μην χάσει η Ευρώπη την ορμή που είχε, την τόσο απαραίτητη σε αυτές τις στιγμές κρίσης, για να μπορέσει να ξαναγυρίσει στην οικονομική και κοινωνική πορεία, τη στεναρή πορεία που ήταν απαραίτητη εκείνη τη στιγμή, το λέω εξορματός όλων μας που εργαστήκαμε τόσο πολύ για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναγνώριση που έχουν εκδηλώσει, έχετε εκδηλώσει έναντι της Ισπανικής Προεδρίας αυτό το εξάμεινο. Όπως είπε και η κυρία Έρτσοκ, πολλές φορές λόγω της κρίσης επισκιάστηκαν οι προσπάθειες της Ισπανικής Προεδρίας, αλλά όποιος καλύζει κάτω από την επιφάνεια της κρίσης έβρισκε τις επιτυχίες της Ισπανικής Προεδρίας. Είναι σημαντικό λοιπόν το ότι έχει αναγνωριστεί αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και πάρα πολύ θετικό ότι υπήρξε η αναγνώριση αυτή, κάτι το οποίο μας ικανοποιεί τα μάλα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τις ευχαριστίες σας. Θα προσπαθήσω τώρα να συνοψίσω την απάντησή μου στα διάφορα ερωτήματα σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την ανάγκη συντονισμού ή τις δυνατότητες συντονισμού για το ηλεκτρονικό ηλεκτρικό συγγνώμη αυτοκίνητο ή το κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να περιμένουν να οριμάσουν τα πράγματα. Εγώ πιστεύω το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τόσο το καθαρά ηλεκτρικό αυτοκίνητο όσο και τα υβριδικά αυτοκίνητα παίζουν κάποιο ρόλο σε αυτή τη στρατηγική. Κάθε χώρα έχει χαράξει τη δική της στρατηγική και εμείς έχουμε τονίσει πάντα η Ισπανική Προεδρία αλλά και η Κομισιόν ότι προωθούμε μια τεχνολογική ουδετερότητα, αλλά και τα ευρεδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δίνουν σημαντικές ευκαιρίες για την τεχνολογική ανάπτυξη της Ευρώπης και γιατί είναι πιο αποδοτικά ηλεκτρονικά, γιατί μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων, αλλά και γιατί οδηγούν στην εξέλιξη νέων τεχνολογιών στον τομέα της αυτοματοποίησης, αλλά και των τηλεπικοινωνιών και στον τομέα του λογισμικού. Όλα αυτά είναι τομείς στους οποίους η Ευρώπη μπορεί να αναλάβει μια ηγετική θέση ως ήπειρος σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή μας ατενίζει. Ο υπόλοιπος κόσμος με μεγάλη προσοχή λόγω της σειράς αποφάσεων που έχουμε λάβει για τα πρώτα μέτρα προώθησης και συντορισμού για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για τα καθαρά αυτοκίνητα. Είμαι πεπισμένο ότι η Κομισιόν όλο και περισσότερο θα επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό συντονισμού, αλλά στο ενδιάμεσο διάστημα εγώ θα ζητούσα από τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν τις προσπαθίες τους. Στην Ισπανία θέσαμε σε κίνηση την ολοκληρωμένη στρατηγική για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με ένα σχέδιο δράση 2010-2012 και βλέπω ότι και άλλες χώρες ακολουθούν παράλληλες γραμμές πλεύσης. Ετέθη το ερώτημα επίσης του κατά πόσο μέσα στο σχέδιο δράσης υπάρχουν κάποιες γραμμές οι οποίες έχουν μεγαλύτερη υψηλότητα, καλύτερα προτεραιότητα για μας. Μία τέτοια γραμμή προτεραιότητος και η οποία δεν είναι προτεραιότητα μονάχα εδώ αλλά και σε άλλους τομείς γιατί ο στόχος μας είναι μια ενιαία αγορά για την ενέργεια, για τα ψηφιακά ζητήματα, μια ενιαία αγορά σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ενιαία αγορά σε όλα τα επίπεδα, αν θέλουμε να έχουμε το απαραίτητο μέγεθος για να έχουμε την κατάλληλη θέση στον κόσμο, χρειαζόμαστε μια τυποποιημένη διαδραστική επιφάνεια για την επαναφόρτιση των ε, ηλεκτρικών αυτοκινήτων που να επιτρέπει και την ε, διαλειτουργικότητα. Επίσης χρειαζόμαστε μηχανισμούς ώστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει επενδύσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα δημιουργία υποδομών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όλα αυτά είναι προαπαιτούμενα. επίση να καλύπτονται οι προδιαγραφές ασφάλειας για να μπορεί να υπάρξει έγκριση κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα αυτά και επίσης σχέδια προώθησης δημιουργίας υποδομών επαναφόρτησης και επανατροφοδοσίας των ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι και τα κρατημέλη και η Κομισιόν θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή ετέθη ένα ερώτημα σε σχέση με την ασφάλεια εφοδιασμού. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια εφοδιασμού. Η Ισπανική Προεδρία έχει αναλάβει μία σειρά από μέτρα, μία σειρά από δράσεις και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό επίπεδο. Για τα εσωτερικά μέτρα ενεκρίθη ο κανονισμός για την κοινοποίηση σχεδίων κάτι το οποίο θα βελτιώσει σίγουρα την, παραχωγή, την παροχή πληροφοριών σε σχέση με τη διαφάνεια των ενεργειακών επενδύσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπάρχει πρόταση κανονισμού για την, τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο, όπου το Κοινοβούλιο έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε επίπεδο πρωτοβουλίες και όπου υπάρχει μια προσωρινή συμφωνία εκκρεμωτήτη της ψήφισης της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την έγκριση της από το Συμβούλιο των Υπουργών. Υπάρχει όμως αυτή η προσωρινή συμφωνία που δείχνει το πόσο έχουμε προχωρήσει στον τομέα αυτό και θέλω και εδώ να ευχαριστήσω αυτά που είπε ο κύριος Τούρμες σε σχέση με τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν από την Ισπανική Προεδρία. για την ασφάλεια και τη μείωση της ενεργητικής εξάρτησης είναι απαραίτητο να δράσουμε και στον τομέα της ζήτησης όσο και στον τομέα της προσφοράς. Για την προσφορά είναι σαφές ότι όλο και περισσότερο αναγνωρίζονται οι ανανεώσιμες ενέργειες ως ασφαλής πηγή ενέργειας και εκμεταλλεύομαι επίσης και το ερώτημα του κυρίου Τέρμς για την μελέτη αυτού του καθηγητή που κατονόμασε σε σχέση με την ε, χρήση των ανανεώσιμων ενεργειών και την απασχόληση. Κάποιος ο οποίος θέλει να έχει μια συνολική μελέτη για τις επιπτώσεις των ανανεώσιμων ενεργειών δεν μπορεί παρά να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν καταστρέφουν θέσει εργασίας. Η καταστροφή θέσεων εργασία οφείλονται στην κατανάλωση πόρων που δεν είναι βιώσιμη και στη δημιουργία στρεβλώσεων. Όταν δηλαδή ακολουθούμε μια οδική γραμμή η οποία δεν βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού της τεχνολογίας. Οι τεχνολογίες και οι ανανεώσιμες ενέργειες μας δίνουν νέες δυνατότητες. Προφανώς θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά τους, να βελτιώσουμε το τεχνολογικό επίπεδό τους. Δεν έχουμε φτάσει στο τελικό λόγο της τεχνολογίας, αλλά ο δρόμος του μέλλοντος, το στίχημα του μέλλοντος έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες ενέργειες. Και λογικά θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή με ένα ευφυή τρόπο. Κατεβρίσαν λοιπόν προσπάθειες από την ε, Ισπανική Προεδρία ώστε η οδηγία που κρίτη το 2009 να αρχίσει να εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη μέσα από τα εθνικά τους σχέδια. Επειδή υπήρχαν και κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με τον καλύτερο τρόπο μεταγραφής αυτής της οδηγίας, διοργανώθηκε αυτό το σεμινάριο υψηλού επίπεδου στην Παμπλώνα τον Απρίλιο που είχε μια μεγάλη επιτυχία λόγω και της παρουσίας εκπροσώπων και της ποιότητας των συζητήσεων. Είμαστε πεπισμένοι ότι στο τέλος όλα αυτά θα δώσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα εθνικά σχέδια τα οποία πρέπει να παρουσιαστούν ως ο νούπο για 30 Ιουνίου θα πρέπει να συνδυαστεί Κομισιόν για να τύχουν περαιτέρω ανάλυση. Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημα που αφορούσε την ενεργειακή εξάρτηση, έχουμε προσπαθήσει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Πήραμε τη σκητάλη από την Σουηδική Προεδρία σε σχέση με την ε, ενεργειακή ετικετοποίηση και την ενεργειακή απόδοση των κτίριων και η Κομισιόν ανακοίνωσε επίσης τη μεταρρύθμιση του σχεδίου ενεργειακής αποδοτικότητας 2010, 2006 μάλλον, κάτι το οποίο προβλεπόταν να γίνει το, τελευταίο, το δεύτερο εξάμεινο του 2009, αλλά καθυστέρησε έκτοτε κατά την άποψή μας και αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί μέσα στο σχέδιο δράσης για την ενέργεια που με τη σειρά του αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το 2020. Η πρόκληση ενώπιον μας λοιπόν είναι να ενσωματώσουμε όλες αυτές τις ψηφίδες σε ένα κοινό παζλ του 2020 και να υπάρξει και η εγκάρσια ε, διασύνδεσή τους με άλλες τεχνολογίες, γιατί βλέπουμε ότι τελικά υπάρχει ένα σύνολο τεχνολογιών που μπορεί να συμβάλλουν σε βελτιώσεις και να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη λοιπόν προς όφελος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προς, προς την ε, ηγετική θέση λοιπόν που μπορούν να έχουν αυτές οι επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και στη συμβολή τους σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ενεργειακή ασφάλεια, την ασφάλεια εφοδιασμού, χωρίς να έχουμε μια Ευρώπη δεόντως διασυνδεδεμένη. Είναι μία από τις προτεραιότητες και ήταν μία από τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας από την αρχή. Αυτό προέρχεται και από την κοινή λογική. Ζητάμε μία κοινή αγορά στο ψηφιακό επίπεδο, μία εναρμόνιση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ζητάμε διαλειτουργικότητα σε κάθε επίπεδο. Θα πρέπει όμως να επιτύχουμε μια Ευρώπη η οποία είναι πιο διασυνδεδεμένη σε ό,τι αφορά την ενέργεια. <clears throat> Αυτός είναι ο βέλτιστος τρόπος δράσης με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ο καλύτερος τρόπος προστασίας της Ευρώπης έναντι κλειδονισμών που οφείλονται σε διακοπή τροφοδοσίας και άλλα προβλήματα ασφάλειας τροφοδοσίας. Στο εξωτερικό επίπεδο Αναφερθήκαμε στις επαφές με τρίτες χώρες. Για το, τα σχέδια της, Ευ... της, της Ενώσεως για τη Μεσόγειο, στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Τη κοινή μας εργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Συμβούλιο Ενέργειας της Ηνωμένες Πολιτείες Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρξε και μία διάσκεψη κορυφής πρωθυπουργών σε περιφερειακό επίπεδο για την ενεργειακή ασφάλεια στη Βουδαπέστη το Φεβρουάριο. Και επανέρχομαι στην Μεσόγειο γιατί το ηλιακό σχέδιο για τη Μεσόγειο ήταν αντικείμενο κάποιας ερώτησης. Συμφωνώ με αυτό που είπε, που ελέγχθη από τους αξιότιμους κύριους βουλευτές, ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο σχέδιο, γιατί πρόκειται για μια περιοχή που μαστίζεται από πολιτικές συγκρούσεις. Αυτός όμως δεν είναι λόγος για να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, κάθε άλλο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας οδηγήσει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας, γιατί πολλές φορές τα πιο δύσκολα και πολιτικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν μέσω συγκεκριμένων προτάσεων δημιουργίας κοινού και αμοιβαίου συμφέροντος για τις χώρες της περιοχής, όπως είναι αυτό το σχέδιο για την ηλιακή ενέργεια αν μπορούμε τώρα να εντοπίσουμε κάποιες χώρες οι οποίες θα ήταν έτοιμες να προχωρήσουν πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση αυτή. Το ίδιο πράγμα που ισχύει και για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια τέτοια εκδοχή. Εγώ νομίζω ότι μέσα στο γενικό πλαίσιο, εάν αναδυθούν τομείς τεχνολογικοί όσο και γεωγραφικές περιοχές όπου μπορεί να υπάρξει ταχύτερη πρόοδος, θα πρέπει να τους ενθαρρύνουμε γιατί μπορεί αυτό να ενθαρρύνει και άλλες χώρες να συνταχθούν με τις χώρες αυτές ή με τους τεχνολογικούς αυτούς τομείς. Μου φάνηκε πολύ εύστοχο το σχόλιο της κυρίας Ερτσόγκ για το συνδυασμό μιας βιομηχανικής πολιτικής, της ψηφιακής ατζέντα και των θεμάτων ενέργειας για να καταλήξουμε σε ένα κοινό τομέα αμοιβαίου εμπλουτισμού και όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εάν προβούμε σε μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνονται οι μεγάλες τεχνολογικές πρόοδοι στον κόσμο και δεν αναφέρομαι τώρα δεν αναφέρομαι στις μεγάλες κλίμακος αλλαγές, αλλά στην δημιουργία καινοτομίας και τεχνολογικής αλλαγής, γίνονται όλα αυτά τα πράγματα από πολλές μικρές εταιρείες, οι οποίες όλες συμπλέουν και συμβάλλουν προς την ίδια αυτή μορφή τεχνολογικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη λοιπόν της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τι τεχνολογίε Όλα αυτά περνάνε από τα χέρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην Ευρώπη εμείς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμα αυτές τις δυνατότητε, δεν έχουμε διερευνήσει πλήρως τον ιστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη σχέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη μεγάλη επιχείρηση και τα κέντρα επίσης δημιουργίας γνώσης που είναι τα πανεπιστήμια. Εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα αναλάβουμε σημαντικά καθήκοντα για να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά αν μπορέσουμε εμείς να ξεκινήσουμε σχέδια όπως αυτά που κάνουμε για να προωθήσουμε την ε, βιομηχανική πολιτική με την ε, αναζωγόνηση της βιομηχανικής πολιτικής και επίσης στον τομέα της ψηφιακής κοινωνίας και τις ενέργειες, νομίζω θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε όλο αυτό τον παραγωγικό ιστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά την Μπέρεκ, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ρίμπικ, η Μπέρεκ μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. σε τομείς όπου θα πρέπει να υπάρξει μια θέση από κοινού αναλύσεων για τις συγκεκριμένες προβληματικές των χωρών μας, πολλές φορές υπάρχει η τάση να τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά σαν να υπάρχει απόλυτη ομοιογένεια μεταξύ των χωρών, κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών είναι σαφές ότι υπάρχει μια πολυμορφία, είναι απαραίτητο να καταλάβουμε από πού έρχεται η κάθε χώρα, ποια είναι τα ισχυρά και αρνητικά στοιχεία της και πού μπορεί να χρειαστεί περισσότερη βοήθεια ή περισσότερο χρόνο. Όλη αυτή η ανάλυση μπορεί να γίνει από τους εθνικούς εκπροσώπους, τους εθνικούς φορείς ε, ρυθμίσεων, που είναι στα πλαίσια της ΜΠΕΡΕΚ, να αναλύσουν από κοινού και να δώσουν στοιχεία μελετών και ανάλυσης ώστε να ληφθούν αποφάσεις από την Κομισιόν. Μου φαίνεται λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να λειτουργήσουν αυτά καλά ώστε να υπάρξει μια επιταχυμένη μετάβαση προς την ενιαία αγορά και να μπορούμε να προωθήσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν πρωτοπόρο ρόλο σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τις αναλύσεις λοιπόν που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τις διάφορες παραμέτρους τεχνολογίας για την κοινωνία της πληροφορίας κτλ. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μικρές και μεσαίες, οι οποίες προεξα... προεξάρχουν σε σημαντικό βαθμό σε ορισμένες περιοχές της κοινωνίας των πληροφοριών. Αυτό το οποίο θέλω να πω λοιπόν είναι ότι αν είμαστε σε θέση να κάνουμε μία επιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επειδή τώρα είναι και η εποχή του Μουντιάλ, να έχουμε ένα είδος ευρωπαϊκής ομάδας, να παίζουμε με τους καλύτερους παίκτες κάθε χώρας και μπορούμε, αν μπορέσουμε να μειώσουμε τις διαφορές μεταξύ των χωρών προς όφελος ενίας αγοράς, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως η περιαγωγή, η δυσκολία να υπάρχουν πολυμερείς άδειες εκμετάλλευσης για τις ε, τηλεπικοινωνίε, να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αν πετύχουμε λοιπόν όλα αυτά από κάθε χώρα να υπάρχει συνεισφορά του καλύτερου και συγχρόνω όλα αυτά να τα συνενώσουμε σε μια ενιαία αγορά, κινούμεθα προ την σωστή κατεύθυνση. Στο τέλο. είναι οι πολίτε, οι χρήστε, οι καταναλωτέ που σε ένα τόσο δυναμικό τομέα μόνο αυτοί μπορούν να επιλέξουν και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να μην μπερδευτούν από την ρευστότητα της των προσφερωμένων τεχνολογιών και ιδεών, είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε λοιπόν και τους πολίτες για ενδεχόμενες καταχρήσεις σε βάρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη ευκαιρία για μένα και χαρά να μπορέσω να μιλήσω μαζί σας και να απαντήσω στα ερωτήματά σας και να παρουσιάσω φυσικά τις επιτυχίες της Ισπανικής Προεδρίας. Και σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Πραγματικά απολαμβάνουμε τις επιτυχίες. Ε, κυρίως στην καθημερινότητά μας είχαμε συνεχώς διαπραγματεύσει με τους συνεργάτες σας, μας βοήθησε πάρα πολύ αυτό και ήταν κάτι το επιτυχές και που μας χαροποίησε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την Προεδρία, ευχαριστήστε και τους υπαλλήλους σας γιατί συνεισέφεραν πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν.